Φίλε uh, Φίλες και φίλοι, ε, καλώς ορίσατε στην δεύτερη, στο δεύτερο τμήμα τη ε, συνεδρίασης της Επιτροπής Απασχολήσεως. Ε, έχουμε κοντά μας προσκεκλημένο ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της, Βουλγαρία, της Βουλγαρικής Δημοκρατίας, κ. Πέτκοφ. Καλώς ήλθατε ε, κύριε Υπουργέ. Σας παρακαλώ να χειροκροτήσετε. Yeah. Ε, and συνεχίζει η πρόεδρος. Είναι μαζί του ο αναπληρωτής υπουργό, σας παρακαλώ να τον υποθετείτε ε, το ίδιο εγκάρδια. Είναι δηλαδή μάλλον η ε, υφυπουργός κυρία Ρουσίνοβα. Αρχίσαμε τη συνεργασία με τους εκπροσώπους της ε, νέας Προεδρίας ήδη από αρκετούς μήνες, γιατί βεβαίως έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Επίσης, έχει διεξαχθεί χθε το βράδυ ήδη ε, τριμερής διάλογος και φτάσαμε μέχρι τα μεσάνυχτα σχεδόν για την οδηγία απόσπασης εργαζομένων. Ήταν ε, η πέμπτη συνάντηση τριμερούς διαλόγου. Βεβαίω δεν μιλήσαμε μόνο για πολιτική, αλλά κάναμε και κάπως παρέα, στο έτσι, διότι με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να εργαστούμε όταν ε, βεβαίως εργαζόμαστε σκληρά για να ε, βρούμε λύσεις μέχρι των ε, διαβουλεύσεων, λύσεις κοινή αποδοχής. Αυτό λοιπόν έγινε χθε το βράδυ. Καλώς ήρθατε λοιπόν και εσείς εκπρόσωποι της κυβερνήσεως και το προσωπικό που σας συνοδεύει. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Υπουργό. Ο κ. Πέτκοφ, όπως είπα είναι υπουργό εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων, για να μπορέσει να κάνει ορισμένες εισαγωγικές παρατηρήσεις. Ορίστε, έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Ουλτσκοκ, αγαπητές και αγαπητοί Ευρωβουλευτές της Επιτροπής ε, Απασχολήσεως. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που εμφανίζομαι ενώπιόν σας για να σας εξηγήσω τις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας και του Συμβουλίου. Επομένως, τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής. Αναλαμβάνει η χώρα μου, η Βουλγαρία, την Προεδρία του Συμβουλίου σε ένα χρονικό σημείο όπου οι Ευρωπαίοι πολίτες αισθάνονται έντονα την ανάγκη να βελτιωθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης αλλά και η κοινωνική προστασία. Χρειάζονται και περισσότερη εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Αντιμετωπίζει το Συμβούλιο σημαντικές προσδοκίες. Εμείς αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη που αναλαμβάνουμε. Οι προτεραιότητες που έχουμε εντοπίσει στον τομέα της απασχολήσεως και κοινωνικής πολιτικής εκφράζουν αυτή την ευθύνη που αισθανόμαστε. Η ενότητα, δικαιοσύνη και πολιτική συνοχής Αυτά τα πράγματα βρίσκονται στην καρδιά του βουλγαρικού οράματος σχετικά με την ανάπτυξη των μηχανισμών που θα χρειαστεί για να καταλήξουμε σε σημαντικά αποτελέσματα στην ε, κοινωνική διάσταση της Ευρώπης. Μέσα στο επόμενο εξάμεινο που θα έχουμε την ε, Προεδρία του Συμβουλίου, η Βουλγαρία θα προσπαθήσει να παίξει τον ρόλο του δίκαιου μισολαβητού. Στην παρούσα φάση του θεσμικού κύκλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα σημαντικό μέρος του θεματολογίου της Προεδρίας μας θα σχετίζεται άμεσα με το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα κλειδιά που βρίσκονται τώρα πια στην φάση των τριμερών διαλόγων. Και σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται να βάλουμε στο κέντρο των ενδιαφερόντων μας τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Έχουμε θετική οικονομική εξέλιξη, οικονομική ανάπτυξη για την ώρα και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε ώστε να βελτιώσουμε την ανθεκτικότητά μας σε μελλοντικέ κρίσεις για να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε απασχόληση, δουλειές δηλαδή και να ενισχύσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη. θα βασιστούμε στα επιτεύγματα των προηγουμένων προεδριών, δηλαδή ιδίω της Εστονικής και ε, κυρίως θα ασχοληθούμε με, το μέλλον της εργασίας, της απασχόλησης θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε προόδους για την επίλυση θεμάτων που έχουν σχέση με την παραγωγική απασχολησιμότητα και μια ε, ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη. Να φέρουμε την προσοχή δηλαδή στις αλλαγές που βλέπουμε στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Θα προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και με βάση βέβαια την κοινωνική καινοτομία. Θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε θέματα ίσων ευκαιριών, μη διακρίσεων και για τον ρόλο των γυναικών στον ψηφιακό κόσμο. Θέλουμε επίσης να εξετάσουμε νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις για πολιτικές απασχόλησης των νέων, καθώς επίσης για μια δίκαιη μετανάστευση και την διασύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης δεξιοτήτων και αναγκών της αγοράς εργασίας. Το μέλλον της εργασίας διασυνδέεται άμεσα και με την επόμενη προτεραιότητα που θα εξηγήσω, δηλαδή τη μελλοντική χρηματοδότηση της κοινωνικής Ευρώπης και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την περίοδο 2014-2020. Εδώ η συζήτηση θα στραφεί γύρω από την περαιτέρω απλούστευση των κανόνων και την στήριξη συνεργειών που θα στοχεύουν σε μια συνοχή οικονομική, κοινωνική και εδαφική. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να παρέχουμε, να βελτιώνουμε μάλλον ευκαιρίες απασχόλησης και τις προσπάθειες για κοινωνική συμπερίληψη και να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε την εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και την διαβίου κατάρτιση υπέρ όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τρίτη μας προτεραιότητα θα είναι να στοχεύσουμε στην προώθηση της έννοιας της ε, ανάπτυξης της παιδικής ηλικίας με ε, ολοκληρωμένες πολιτικές, με ασφαλή υποστήριξη των οικογενειών για ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά τους. Πρόκειται δηλαδή για επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό. Η τέταρτη προτεραιότητά μας θα είναι η ενασχόληση με τους ανθρώπους που έχουν αναπηρίες. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και ελευθερίες χωρίς καμιά διάκριση. Αυτό μάλιστα περιλαμβάνεται και σε αριθμό στρατηγικών εγγράφων και στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι αναγκαίο να προωθηθεί και να γίνει πιο συγκεκριμένη η ε, προσέγγιση αυτή ώστε να παρασχεθούν και να είναι εγγυημένα τα ίσα δικαιώματα για τους αναπήρους. Αυτή θα είναι η προσπάθειά μας και θα κάνουμε και κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρώσουμε τον τριμερή διάλογο για την για την νομοθεσία για την προσβασιμότητα από την άποψη των ε, αναπήρων προσώπων. Το ίδιο για τα δικαιώματα των εργαζομένων, χωρίς βεβαίως να μειωθεί η δυνατότητα των επιχειρήσεων να παρέχουν υπηρεσίες. Θα δώσουμε ε, τελική μορφή στις συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την οδηγία απόσπαση εργαζομένων. Θα συνεργαστούμε μαζί σας προς την κατεύθυνση μιας συνολικότερης προσέγγισης για τα δύο τελευταία κεφάλαια της πρότασης αναθεώρησης του κανονισμού 883, δηλαδή για επιδόματα ανεργίας και για, για ε, προσωρινές διατάξεις. Ιδιαίτερη ε, σημασία θα αποδώσουμε στην ε, ασφάλεια της υγείας και στην ασφάλεια στις, στους τόπους εργασίας για την προστασία των εργαζομένων και απέναντι σε καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες. Θα συνεχίσουμε δε και την προσπάθεια στους κανονισμούς για τους οργανισμούς SEDEFOP, EU, OSA και Eurofound. Στο τέλος της σύντομης αυτής ομιλίας επιτρέψτε μου να επανέλθω σε ένα στοιχείο που θα είναι το κλειδί, στην καρδιά των προσπαθειών μας. Ενώ τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα υπάρξει διαθεσμική διακήρυξη, μάλλον υπήρξε, η οποία ήδη υπογράφηκε στο Γκέτεμποργκ για ε, τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για την εφαρμογή της ήδη από τώρα και στο επόμενο εξάμεινο με τις σχετικές πρωτοβουλίες στη δέσμη μέτρων κοινωνικής δικαιοσύνης. Θα εργαστούμε ενεργά και για άλλες νομοθετικές προτάσεις οι οποίες συνδέονται άμεσα με την βελτίωση των συνθήκων εργασίας των Ευρωπαίων πολιτών καθώς και την βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ο νέος κύκλος Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και η ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων και το σχετικό θεματολόγιο θα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στις δύο συναντήσεις του ε, Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ, δηλαδή Απασχόλησης Κοινωνικής Πολιτικής Υγείας και ε, Καταναλωτών. Αυτά θα γίνουν τον Μάρτιο και Ιούνιο του 2018. Είμαι βέβαιος ότι το σύνθημα της Βουλευτικής Προεδρίας στα αγγλικά United we stand strong, δηλαδή όλοι ενωμένοι, θα είναι και το κλειδί για την επιτυχία μας στον χώρο της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής. Μέσα στο επόμενο εξάμεινο θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εφαρμοστεί αυτό. Ενωμένοι θα αποδειχθούμε ισχυροί και ικανοί να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή άλλη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, λέει ο Πρόεδρος και μήπως η κυρία Ρωσινόβα θέλει να προσθέσει κάτι Όχι, καλώς. Μπορούμε να θέσουμε ερωτήσει όμως και στους δυο σας, έτσι δεν είναι. Ωραία. Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Θα καλέσω πρώτα τους ε, συντονιστές των πολιτικών ομάδων να θέσουν ερωτήσεις. Τα άλλα μέλη πλην συντονιστών μπορούν να ζητήσουν να λάβουν τον λόγο. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον συντονιστή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κύριο Κάσα. Ορίστε κύριε Κάσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τον Υπουργό και την Υφυπουργό που ήρθαν να παρουσιάσουν τις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας. Ε, πολύ χαίρομαι για αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα της Βουλγαρικής Προεδρίας που περιλαμβάνει πολλά θέματα κοινωνικής πολιτικής και είμαι σίγουρος ότι η Προεδρία είναι καλά προετοιμασμένη για να πετύχει τους στόχους της. Μέσα σε έξι μήνες θα καταφέρει όσο μπορεί περισσότερα. Η Προεδρία βέβαια έρχεται στα πλαίσια δύο πολύ σημαντικών ε, συζητήσεων που είναι το Brexit και το πολιτές δημοσιονομικό πολιτές δημοσιονομικής προοπτικές που πιθανόν επισκιάσουν άλλες προτεραιότητες της ε, Βουλγαρικής Προεδρίας. Με ενδιαφέρει πολύ και θα έχουμε την έκθεση αυτή όσον αφορά ε, τη φροντίδα των ε, παιδιών, τους γονείς που φροντίζουν τα παιδιά. και είναι κάτι που είναι του πρώτου πυλώνα, κοινωνικά δικαιώματα. Συζητιέται ήδη, όπως γνωρίζουμε, στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι ερωτήσεις μου έχουν ως εξή. Θέλουμε να ξέρουμε τα σχέδια και τις φιλοδεξίες της Βουλγαρικής Προεδρίας για αυτή τη σημαντική υπόθεση και δεύτερον, ποιοι είναι οι τομείς όπου η Προεδρία περιμένει να αντιμετωπίσει περισσότερες δυσκολίες από ό,τι αλλού. Ευχαριστούμε κύριε Κάσα, λέει πρόεδρος. Συνεχίζουμε με την κυρία Γιονγκέριους που είναι συντονίστρια των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για την παρουσία σας. Πράγματι, είσαστε μια πρωτιά, έτσι, γιατί είναι η πρώτη φορά που έχει η Βουλγαρία την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα σε μια πολύ σημαντική στιγμή, όχι μόνο για τα θέματα που έθιξε ο συνάδελφος Κάσα, αλλά επιπλέον επειδή αν ε, θέλουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας έγκαιρα στα πλαίσια αυτής της θητείας, θα έλεγα ότι εσείς είσαστε η τελευταία μας ευκαιρία για να τα καταφέρουμε. Πράγματι, χτες αρχίσαμε τι συζητήσει τριμερή διάλογο για την απόσπαση των εργαζομένων. Γιατί είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση και σας ευχαριστώ πολύ για το έργο σας από αυτού. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με δύο πράγματα. Πρώτον, στις προτεραιότητές σας Μιλάτε για τα παιδιά και την ένδια από την οποία υποφέρουν τα παιδιά. Δεν θα πρέπει να περιμένω τη στήριξή σας για κάτι που ήδη προωθεί η ομάδα μας εδώ και πολύ καιρό και που είναι μια εγγύηση για τα παιδιά προκειμένου κανένα παιδί στην Ευρώπη να μην υποφέρει από φτώχεια, να μην μεγαλώνει μέσα στη φτώχεια. Δεύτερον, για κάτι στο οποίο επίσης αναφέρθηκε ο συνάδελφος Κάσα. Τι πιθανότητες έχετε, πιστεύετε, να πετύχετε γενική συμφωνία για την ισορροπία αυτή ε, ζωής και εργασίας. Είναι και αυτό σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. είναι ένα θέμα που βρίσκεται ψηλά στις δικές μας προτεραιότητες και γιατί έχουμε κακή εμπειρία από τις προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε με το Συμβούλιο όσον αφορά την οδηγία για την ε, μητρική άδεια. Οπότε ελπίζω μόλις τελειώσει την έκθεσή του κ. Κάσα να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τριμερή διάλογο και από αυτού. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Και συνεχίζουμε με το συντονιστή από το ECR. Η κυρία Μάκεντάιρ δεν είναι όμως εδώ. Κάποιος την αντικαθιστά. Όχι. Περνάμε στους φιλελεύθερους, Άλτε, αλλά δεν βλέπω τον κύριο Καλβέρ Σαμπού. Ούτε κυρία Λαβάτζοβα. Γκουε, NGL, ούτε. Από Πιμέντα Λόπες, όχι. Πράσινη. Ναι. Η κυρία Λάμπερτς. Παρακαλώ, κυρία Λάμπερτς. Ευχαριστώ και εγώ του υπουργού που είναι παρόντες εδώ σήμερα. Καλώς ήρθατε η εμπειρία μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολλών από εμά, είναι ότι οι προεδρίες των ε, μικρών χωρών συχνά είναι πολύ πιο δυναμικές και δημιουργικές και καταφέρνουν να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα στο Συμβούλιο από ότι οι μεγάλες καταφέρνουν να μετακινήσουν το Συμβούλιο από τις θέσεις του και να πετύχουν οι διαπραγματεύσεις. Ελπίζω αυτή να είναι και η στάση της δικιά σας ε, Προεδρία και αυτό να κάνετε κι εσείς στους τριμερείς διαλόγους στους οποίους συμμετέχετε. Ένα ζήτημα για την μπλε κάρτα. Μιλήσαμε για μια δίκαια πολιτική μετανάστευσης. Αυτή η μπλε κάρτα προς το παρόν αντιμετωπίζει εμπόδια. Μέχρι τώρα έχουμε δει να υπάρχουν εντάσεις ανάμεσα στα Υπουργεία Εσωτερικών που βλέπουν να πρόκειται πώς να το πω, έχουν πολύ σκληρές και αυστηρές απόψεις για τη μετανάστευση, ενώ υπάρχουν άλλοι υπουργοί καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα, οι υπουργοί εργασία δηλαδή, καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα ότι μας χρειάζονται δεξιότητες και από μέρη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι αγνοούμε τις δεξιότητες που έχουμε στο εσωτερικό μας. Λοιπόν, εσείς πώς το βλέπετε αυτό. Οι Υπουργοί Εργασίας πιστεύετε να μπορέσουν να επηρεάσουν περισσότερο τα πράγματα της διαπραγματεύσεις για την μπλε κάρτα, προκειμένου να υπάρχει μια πιο θετική στάση. Και τώρα για τις νέες ε, προτάσεις όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Προς το παρόν μας απασχολεί πολύ ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η νομοθεσία. Μια τέτοια αρχή έπρεπε να υπάρχει εδώ και καιρό. Οπότε αναρωτιέμαι κατά πόσο εσείς πρόκειται να το προθήσετε αυτό το θέμα πιο γρήγορα έτσι όπως θα θέλαμε κι εμείς. Πρόεδρο, ευχαριστούμε από το ENF, ο κύριος Μαρτάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Πετκόφ που είναι της, ε, των που είναι και δικιά μας αρμοδιότητα και την Υφυπουργό. Μερικές ομάδες, και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, δεν είναι παρούσες εδώ. Και έτσι δεν έχουν την ευκαιρία να σας ρωτήσουν πράγματα. Εν υπάρχει η, ο χάρτης πορείας Μιλήσαμε για την εκπαίδευση, την κατάρτιση για τα παιδιά, τους γονείς, τους εργαζόμενους, τους απασπασμένους, στο τριμερή διάλογο για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, για τον κοινωνικό και ευρωπαϊκό πυλώνα. Όλα αυτά που μας είπατε, κατάλαβα ότι έχουν συμφωνηθεί και γι' αυτό και μας τα λέτε. Όμως εγώ σας συγχαίρω για την πρώτη συνεδρίαση χτες βράδυ του τριμερούς διαλόγου, αργά τη νύχτα. Είχατε την τόλμη, το θράσος θα μπορούσα να πω ακόμα, να θέσετε τα πιο λεπτά σημεία. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στα θέματα αυτά τα μεγάλα που εσείς θέλετε να προωθήσετε μέσα στο επόμενο εξάμεινο. Ανάπτυξη της σχέσης της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς. Είναι κάτι για το οποίο μιλάμε, ξαναμιλάμε, ξαναξαναμιλάμε, αλλά κανείς δεν βρίσκει τη λύση. Πώς θα έχουμε πρόσβαση στην καινοτομία, πώς θα έχουμε την κοινωνική συνοχή μέσω της άτυπης μάθησης, όχι μόνο της επίσημης, της τοπικής. Τώρα το 2017 με το τρίο των ε, προεδριών είχαμε αναφερθεί στη στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις startup προκειμένου να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαφορετικού είδους χρηματοδότηση. Ακόμα και στη Γαλλία όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι οι μικρομεσαίες που δημιουργούν το 90% των θέσεων απασχόλησης και όχι οι άλλες, οι μεγάλες που θέλουν να μας επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες. Τώρα η ερώτησή μου που μπορεί βέβαια να σας ανοχλήσει λίγο. Είσαστε υπουργός της Βουλγαρίας, στηρίζετε τη Βουλγαρία και καλά κάνετε. Ρωτάω, είσαστε ικανοποιημένο από αυτό το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως τι λέτε και αυτές τις μικρές χώρες στη γειτονιά σας που θέλουν να εντεχθούν τους αφήνουμε τη θέση να ενταχθούν με τις δικές τους εσωτερικές ε, πεπιθήσεις, όπως στη δικιά σας την περίπτωση, πρώτα η Βουλγαρία. La Bulgarie d'abord. Αυτό ήταν ο πρώτος γύρος ερωτήσεων. Και θα έχουμε και άλλες ερωτήσεις μετά. Μην ανησυχείτε. Οπότε παρακαλώ για να απαντήσετε Ευχαριστώ πολύ για τα θερμά σας λόγια, τη θερμή σας υποδοχή και τις ερωτήσεις σας. Επιβεβαιώνω για άλλη μια φορά ότι οι προτεραιότητες του Συμβουλίου είναι και προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σας απασχόλησης. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στον κύριο Κάσα και την κυρία Γιουγκέριους πρώτα. για την ισορροπία, την οδηγία αυτή δηλαδή, για την ισορροπία προσωπικής και εργασιακής ζωής. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Είναι πρώτη προτεραιότητα για τη δικιά μας την Προεδρία. Και η φιλοδοξία μας είναι να έχουμε μια κοινή προσέγγιση στο Συμβούλιο. Το Μάρτιο που θα έχουμε την πρώτη συνάντηση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Που αποτελεί μέρος του κοινωνικού πυλώνα. Γνωρίζουμε ότι οι χώρες μέλη στηρίζουν τους στόχους της οδηγίας αυτής. Και γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε συμφωνία, όπως και σε άλλα θέματα. για την αμοιβόμενη γονική άδεια. Μην ξεχνάμε όμως ότι όλες οι χώρες έχουν τις δικές τους ξεχωριστές παραδόσεις και απαιτήσεις. Οπότε πρέπει πολύ προσεκτικά να προσεγγίσουμε το θέμα. Και έτσι όπως το κάνουμε εμείς, πιστεύω θα βοηθήσει να πετύχουμε τελικά συμφωνία στο Συμβούλιο. αλλά τονίζω ότι αποτελεί προτεραιότητα της Βουλγαρικής Προεδρίας. Και ελπίζουμε και εμείς να πετύχουμε τους στόχους αυτούς που σας περιέγραψα. Μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας επίσης έχει να κάνει με, την, με τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, στο ανθρώπινο κεφάλαιο για τα παιδιά, ε, στήριξη της οικογένειας. Είναι μια προσέγγιση στραμμένη στο μέλλον. Που σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα διάφορα στάδια ανάπτυξης της ε, ζωής. Και το υψηλό επίπεδο φτώχειας που πλήττει τα παιδιά είναι κάτι που πρέπει να έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας και να το λύσουμε. Έρχομαι τώρα στην ερώτησή σας για την μπλε κάρτα. Πιστεύω ότι ρόλος των ε, Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικών Θεμάτων και Απασχόλησης είναι πολύ σημαντικός και η συμμετοχή τους είναι αναγκαία. Θα βγάλουμε από το ψυγείο λοιπόν το θέμα. Διότι εφόσον υπάρχουν νόμιμοι οδοί, νόμιμη πρόσβαση πολιτών τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. και θα δώσει δυνατότητα απασχόλησης με τη χρήση ακριβώς της μπλε κάρτας και θα μπορέσουν έτσι άνθρωποι με υψηλά προσόντα και δεξιότητες να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει την οικονομία μας, θα αποτελέσει άλλη μια πηγή για την οικονομία μας. Ελπίζω λοιπόν να προχωρήσουμε και σε αυτό το θέμα. Τώρα, πώς θα δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για την ε, κινητικότητα στην εργασία. Θέλουμε να δημιουργηθεί αυτή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εργασίας. Είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρχές Μαρτίου θα έχω περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει αυτή την αρχή. Αν μας πει περισσότερα η Επιτροπή αρχές Μαρτίου, θα συμπεριλάβουμε αυτό το θέμα στο πρώτο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων το Μάρτιο. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί τέτοιες πρωτοβουλίες βοηθούν στην εφαρμογή των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αναφέρθηκα σε αυτό στην αρχή όταν αναφέρθηκα στις προτεραιότητές μας. Χαίρομαι που λέτε ότι χτες το βράδυ ήταν καλή η παρουσία μας και η δουλειά μας. Αυτή είναι η αποστολή μας και να ξέρετε ότι θα συνεχίσουμε το τόσο καλό έργο που επετέλεσε η Εστονική Προεδρία. <clears throat> θα προσπαθήσουμε στη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας να κλείσει αυτή η υπόθεση. Είναι μια φιλοδοξία που έχουμε και συνεχίζουμε να έχουμε και θα έχουμε και στον επόμενο τριμερή διάλογο. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο προστατεύει τους εργαζόμενους, χωρίς να περιορίζει όμως την ελευθερία παροχής υπηρεσιών μέσα στην ενιαία αγορά. Συμφωνώ επίσης με τον κύριο Μαρτά για την σχέση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Αυτή η σχέση είναι πολύ σημαντική. Αλλάζουν συνεχώς οι συνθήκες. Ε, χρειάζεται ένα σύστημα εκπαίδευσης και επαγγελματική εκπαίδευσης με ιδιαίτερο δυναμισμό για να ανταποκριθεί στις αλλαγές αυτές. Τώρα είπα ήδη ότι θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στις δεξιότητες που είναι αναγκαίες σε μια σύγχρονη αγορά εργασίας. Και ένα από τα πράγματα που σκοπεύουμε να κάνουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας είναι ότι θα εγκρίνουμε σύσταση για την μαθητεία, που είναι πολύ σημαντικό προκειμένου ακριβώς να προσαρμόζονται οι νέοι στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, apprenticeship. Η Βουλγαρία είναι μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 10 χρόνια και για πρώτη φορά αναλαμβάνουμε την Προεδρία στο Συμβούλιο. Εκ μέρους λοιπόν του Συμβουλίου μπορώ να πω ότι ναι και οι μικρές χώρες τελικά έχουν τη θέση τους σε αυτή τη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να περάσουμε απευθείας στον επόμενο κύριο μιλητών με τον κύριο Κόζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον Υπουργό για το φιλόδοξο πρόγραμμα της Βουλγαρικής Προεδρίας. Έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Μιλήσατε για ανθρώπους με αναπηρίες. Εδώ στην Επιτροπή Απασχόλησης είχα αναλάβει ως εισηγητής το, τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα. Και έχουμε συναντηθεί πολλές φορές με εκπροσώπους του Συμβουλίου από τις διάφορες προεδρίες ε, εν ώψη των τριμερών διαλόγων. Ελπίζω ότι αυτό θα μας οδηγήσει σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι αποδεκτό από όλους. Οι πολίτες με αναπηρία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ελπίζω ότι θα είναι ικανοποιημένοι με την νέα νομοθεσία. Η ερώτησή μου όμως είναι ποια η θέση της Βουλγαρικής Προεδρίας ως προς την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναφέρει ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν υποδομές μεταφορών, οχήματα, συγκοινωνίες, τουρισμός και σχετικές υπηρεσίες όπου να προβλέπεται πρόσβαση ε, με, ε, για τους ανθρώπους με αναπηρίες και για τους τομείς που δεν προβλέπονται στην αρχική πρόταση. Υπάρχει περίπτωση για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει αυτή τη θέση. Ήθελα να γνωρίσω και τη δική σας άποψη. Ευχαριστώ. Υπουργέ, θέλετε να ξεκινήσετε την απάντησή σας σε αυτό. Όχι, να ακούσουμε και μια δεύτερη ερώτηση, ο κύριος Νόβακοφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προτιμήσω να μιλήσω βουλγαρικά. Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας και τις διευκρινήσεις που μόλις μας δώσατε. Ως εκπρόσωπος μιας από τις μεγαλύτερες χώρες των Βαλκανίων, θα ήταν καλό να μας πείτε ποια είναι και η θέση σας για κάποια ζωτική σημασία θέματα και φακέλους που θα εξεταστούν και θα αναθεωρηθούν τα ερχόμενα χρόνια. Εγώ ασχολούμαι με τα ευρωπαϊκά ταμεία και τη λειτουργία του ευρωπαϊκού προπολογισμού, τι προπτικέ του δηλαδή, ω το 2020. Ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σα για τα χρηματοδοτικά εργαλεία τη Ένωση. Σε ό,τι αφορά όμω τον κοινωνικό τομέα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, την εγγύηση για του νέου, το Ταμείο Προσαρμογή ε, στην παγκοσμιοποίηση. Καθώς, καθότι γνωρίζω ότι τα τελευταία χρόνια στη Βουλγαρία έχουν βοηθήσει πάνω από 60.000 νέους στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχουν βρει δουλειά ε, αυτοί οι άνθρωποι. Πώς σκοπεύετε να εκμεταλλευτείτε αυτήν την όθηση που έχει δοθεί και να βεβαιωθείτε ότι προσφέρετε εργασία σε όσο το δυνατόν περισσότερους νέους, στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Να ακούσουμε και μια τρίτη ερώτηση. Μάλιστα, κυρία Τόμτς. Ευχαριστούμε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε για την ομιλία σας και για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων. Νομίζω έχετε επιλέξει κέρια ζητήματα. Ήδη όμως έχουν τεθεί τα σημαντικότερα ερωτήματα από τους συναδέλφους. Εγώ έχω μία επιπλέον ερώτηση. Αφορά ένα πολύ επίκαιρο θέμα που μας έχει απασχολήσει και όλες τις τελευταίες ημέρες. Η νέα κυβέρνηση της Αυστρίας έχει ε, προτείνει την, ε, τον υπολογισμό του επιδόματος για παιδιά με βάση αυτό που ισχύει σε χώρες προέλευσης. Δηλαδή να υπάρξει ενός είδου ε, τιμαριθμική, προσαρμογή του επιδόματος. Αυτό όμω δεν συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία για τα κοινωνικά συστήματα. Πώς σκοπεύετε να το επιλύσετε στο μέλλον. Εδώ πιστεύω ότι έχετε να διδραματίσετε έναν ρόλο. Έχετε να λάβετε μια σημαντική απόφαση για ένα σημαντικό θέμα. Αυτό το θέμα δηλαδή. Ε, και επόμενη ερώτηση. σκοπεύετε να έχετε ενεργό ρόλο σε αυτές τις συζητήσεις. Και τον κανονισμό 883 του 2004. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι και προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Благодаря за зададените въпроси. Ако ми позволите да Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας, ξεκινώντας από την κυρία Τόντ. Ε, σε σχέση με την ε, αναθεώρηση του κανονισμού 883 του 2004 για το συντονισμό των ε, συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Βεβαίως, χρειάζεται να ενημερώσουμε τα κοινωνικά μας συστήματα και να βεβαιωθούμε ότι η προστασία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επαρκής. Αλλά μια και το αναφέρω αυτό, να θυμίσω ότι μια από τι προτεραιότητε τη Βουλγαρική Προεδρία είναι ακριβώ να υπάρξει μια εν μέρη γενική προσέγγιση για τα τελευταία κεφάλαια του κανονισμού αυτού, του 883, κεφάλαια τα οποία ακριβώ έχουν να κάνουν με τα επιδόματα για τους εργαζομένους και τις πρόσθετες διατάξει. Δεν σκοπεύουμε να επιστρέψουμε σε κεφάλαια τα οποία έχουν κλείσει και μια εν μέρη γενική προσέγγιση έχει ήδη συμφωνηθεί στα κεφάλαια αυτά. Να θυμίσω ότι στο τελευταίο Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων του Δεκεμβρίου η εν μέρη γενική προσέγγιση συμφωνήθηκε για δύο τουλάχιστον κεφάλαια από αυτόν τον κανονισμό. Ο σκοπός μας θα είναι εντός τη βουλγαρικής προεδρία να συμφωνήσουμε μια εν μέρη γενική προσέγγιση για τα επιδόματα ενεργείας και τις ε, επιπρόσθετες διατάξεις. Δηλαδή, σκοπεύουμε να εργαστούμε συστηματικά για να προωθήσουμε το φάκελο αυτό μαζί με την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Είναι σημαντικά και τα δύο για να διασφαλίσουμε τα εργασιακά δικαιώματα των πολιτών. Επίσης, ε, το ίδιο και η παροχή υπηρεσιών στην ενιαία αγορά. Τώρα για την ερώτηση του κ. Νόβακοφ. Εντός της Βουλγαρικής Προεδρίας σκοπεύουμε να θέσουμε το ερώτημα για το ποιο θα είναι το μέλλον της κοινωνικής Ευρώπης και την χρηματοδότησή της πιο συγκεκριμένα. Μετά το σημερινό μάλιστα πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που λύγει το 2020. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Νομίζω είναι σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι τα κονδύλια φτάνουν στα χέρια των πολιτών ευκολότερα. Θέλουμε να διευκολυνθούν οι πολίτες στην πρόσβασή τους. Θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια. Αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε σχέσεις συνεργασίας και θα μπορέσουν ενδεχομένως να φτάσουν και στο στόχο τους τα κονδύλια, να ταπανηθούν για το σωστό σκοπό. Εντό του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και στη διάρκεια τη Προεδρία μα θα κοιτάξουμε ακριβώ και τη χρηματοδότηση της, ε, της πηγές χρηματοδότησης της κοινωνικής Ευρώπης. Ακόμη και για το διάστημα μετά από αυτήν την περίοδο. Αυτό αφορά και την ερώτησή σα για τα χρηματοδοτικά εργαλεία ανέφερε ότι μια από τις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας στον τομέα των εργασιακών δικαιωμάτων και των κοινωνικών πολιτικών θα είναι ακριβώς οι άνθρωποι με τις αναπηρίες και η προστασία των δικαιωμάτων τους, καθώς και η προσφορά ε, τέτοιων προποθέσεων σε αυτούς τους πολίτες, ώστε να μπορούν να εξασκούν τα δικαιώματα και να απολαμβάνουν τις ελευθερίες τους. Ε, υπ' αυτήν την έννοια, η προτεραιότητά μας είναι να ολοκληρώσουμε επιτυχώς τον τριμερή διάλογο για την ε, νομοθεσία σχετικά με την ε, κοινωνική πρόσβαση. Είχαμε τουλάχιστον δύο συναντήσεις ε, στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου και αρκετές τεχνικές συνεδριάσεις. Προσπαθούμε να καλύψουμε όλα τα σημεία που αφορούν την πράξη αυτή για την πρόσβαση των ανθρώπων με αναπηρίες και σημειώνουμε την παρατήρηση του Ευρωκοινοβουλίου για την διεύρυνση του πεδίου του κανονισμού. Για μα είναι σημαντικό το ζήτημα αυτό, ο φάκελο να περατωθεί εντό τη ε, της Προεδρίας μας. Είναι μια από τι προτεραιότητέ μα οι πολίτες με αναπηρίε. Μάλιστα επαφιόμαστε στην δική σας την υποστήριξη και συνεργασία και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων ανυπομονούμε για την ε, ε, συνεργασία μας και με το Κοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα δύο σημαντικά αυτά ζητήματα. Ευχαριστώ. Να προχωρήσουμε. Ο κύριος Πυρίνσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, κυρίες Υπουργέ, χαίρομαι πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Ε, χαρήκαμε που ακούσαμε τις δικές σας απόψεις και τις προτεραιότητές σας για το εξάμεινο της Βουλγαρικής Προεδρίας, ιδίως για τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας αυτή εδώ την Επιτροπή. Κάποιος ανέφερε τα μικρότερα κράτη-μέλη και το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν. Νομίζω ότι υπό τις δεδομένες συνθήκες εμείς έχουμε να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στη δουλειά της Ευρώπης. Γνωρίζουμε πολύ καλά το τι προκλήσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως μικρά κράτη-μέλη. Αυτά ε, τα κράτη έχουν κάποιες φορές ιδιαίτερα προβλήματα ως μικρότερα κράτη, αλλά πρέπει να τα δουν υπό την οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Ε, επίσης είναι σημαντικό ε, ότι η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια με την κρίση που ξεκίνησε το 2008 με μια μικρά περίοδο λιτότητας περνάει τώρα σε μια περίοδο ανάκαμψης. αναθέρμανσης της οικονομίας. Όμως υπάρχει και ένα διάχυτο άγχος, διότι την ανάπτυξη δεν την απολαμβάνουμε τον ίδιο τρόπο όλα τα κοινωνικά στρώματα. Χθε μόλις το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στον Ταβός, ε, ανέφερε στην ομιλία της ακριβώς αυτό το πρόβλημα, ότι η οικονομική αύξηση η παραγωγή περισσότερου πλούτου δεν διανέμεται δικαίως και ισότιμα. Κάποιες φορές μάλιστα εντείνει τις ανισότητες. Αυτό με φέρνει ακριβώς και πάλι στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Δεν προέκυψε κατά τύχη. Ήταν μια έκφραση μια χειροπιαστή έκφραση αυτού του διάχυτου άγχου που έχουμε αφουγκραστεί και αισθανθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Ήταν ένα μικρό βήμα, αλλά εάν ε, ο κοινωνικό κατάλογο προτεραιοτήτων δεν συμπεριληφθεί στην ατζέντα μα, θα υποστούμε δυσμενεί συνέπειε. Θα πάω κάτι, πίσω σε κάτι που ανέφερε ο κύριος Μαρτά. Ε, το κατά πόσον ε, απογοητευτήκαμε ε, ως Βουλγαρία από την ε, προσχώρησή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι και μήπως τώρα πρέπει να αρχίσουμε να προασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας. Η διάθεση που επικρατεί στη Βουλγαρία και η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι τα βουλγαρικά συμφέροντα καλό είναι να τα προσπιστεί κανείς στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συνδυάζοντάς τα με, την, με αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή θέλουμε η Ευρώπη να γίνει μια ανταγωνιστική γεωγραφική περιοχή. Μια ανταγωνιστική ήπειρος. Και έχοντας ε, αυτά τα στοιχεία κατά νου, πιστεύω ότι η δική σας Προεδρία, ιδίω στον τομέα των κοινωνικών δικαιωμάτων και της απασχόλησης, μπορεί να ε, προσφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Ε, τώρα κάποιες ερωτήσεις. Τα ρώτησαν και η κυρία Γιουγκέριους και ο κύριος Κάζα για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου. Αυτό πραγματικά θα ένα πολύ καλό τεστ, μια πολύ καλή δοκιμασία για να δούμε πώς οι σχετικές διατάξεις του κοινωνικού πυλώνα μπορούν και θα εφαρμοστούν. Οπότε η ερώτησή μου είναι λίγο αφηρημένη, λίγο θεωρητική από αυτήν την έννοια. Ο κύριος Κάζα ανέφερε τις πιο περίπλοκες πτυχές του θέματος, του φακέλου αυτού, ε, εδώ υπάρχει ένα θέμα αρχής που πρέπει να συζητήσουμε. Και έχει να κάνει με το εξής. Οι διατάξεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιλύουν το θέμα, το πρόβλημα της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ίσα ίσα η διάθεση που έχει επικρατήσει είναι ότι αυτές οι διατάξεις θα γύρουν περισσότερα εμπόδια. Επίσης, πιστεύει ο κόσμος ότι το σύστημα που προτείνεται δεν θα αξίζει τον κόπο και δεν θα αξίζει να χρηματοδοτηθεί, διότι θα αναστείλει την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών υπερασπιζόμαστε την αντίθετη άποψη. Εμεί θέλουμε ένα εξισορροπημένο σύστημα με ισότιμη κατανομή των ε, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εντό μια οικογένεια. και επιπλέον ευκαιρίες φροντίδας των ηλικιωμένων της τρίτης ηλικίας. Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο θα επιτρέψει να υπάρχει ακόμη καλύτερη ανταγωνιστικότητα και δυνατότητα για ανταγωνισμό των εταιριών. Υπ' αυτήν την έννοια, οι κοινωνικοί εταίροι και οι συλλογικέ συμβάσει θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Προσπαθώ εδώ να είμαι τελείω ψυχρός και αντικειμενικός. Γι' αυτό θα ρωτήσω το εξή. Τι χρονοδιάγραμμα προτείνετε για αυτές τις συζητήσει εσείς. Και επιπλέον έχω μία πρόταση Μία προτροπή να σας κάνω. Θα ηγηθείτε στο εξάμεινο της Βουλγαρικής Προεδρίας ε, στις συζητήσεις των, θέματων, των θεμάτων αυτών. Θα τις διευθύνετε εσείς. να μην ξεχνάμε τι διεθνεί συνθήκες για τα θέματα αυτά, διότι δεν κατοπτρίζουν το κοινωνικό πρόσωπο που η Ευρώπη θέλει να καλλιεργήσει. Τα τελευταία χρόνια το θέμα ήταν ότι έμεινε στα μετόπιστα η κοινωνική Ευρώπη, διότι κοιτάζαμε να προωθήσουμε την χρηματοοικονομική σταθεροποίηση. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό, διότι αναπόφευκτα το όλο θέμα θα χρειαστεί να το εξετάσετε. Ως προς την εγγύηση για τα παιδιά, η ομάδα μας θεωρεί το θέμα αυτό ως προτεραιότητα. Η αύξηση της ένδυας ε, στην ηλικία την παιδική και οι τάσεις που έχουν δημιουργηθεί, 26,4% πολιτών κάτω των 17 να κινδυνεύουν να περιέλθουν σε συνθήκες φτώχειας. Το πρόβλημα στη Βουλγαρία είναι διπλάσιο από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Βλέπω ότι η κυρία Ουλφσκοκ ήδη γνέφει αλλά μάλλον θα με προσκαλέσει να ολοκληρώσω. Είχα και άλλες ερωτήσεις να θέσω, αλλά μία μόνο θα μου επιτρέψω και μετά θα πάυσω. Ε, ο Οργανισμός Εποπτείας της Απασχόλησης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εποπτείας, είπατε ότι θα συζητηθεί τον Μάρτιο είναι ένα θέμα ε, αποφασιστικής σημασίας για τα θέματα απασχόλησης που είναι και η σφαίρα των αρμοδιοτήτων σας. Ήθελα να σας καλέσω να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για την παράνομη και αδήλωτη εργασία. Ε, πέρσι, στα τέλη της χρονιάς, διοργανώθηκε μια ακρόαση στην Επιτροπή αυτή. Ήρθαν εδώ εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής της πλατφόρμας και διάφοροι υπεύθυνοι από κοινωνικές υπηρεσίες της Ευρώπης. Εξεπλάγησαν οι συνάδελφοι που άκουσαν να γίνονται έντονες συζητήσεις και να υπάρχουν έντονες τυχομηθίες για το όλο θέμα. Ε, η όλη η εμπειρία βρίσκω ότι ήταν πολύτιμη αξιολογία και θα μπορούσατε να την ε, αξιοποιήσετε κι εσείς. Εν τέλει να πω ότι το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο συμπεριλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις ε, πολλέ ιδέε για το τι θα γίνει την περίοδο μετά το 2020. Εκεί προτείνεται και μια ιδέα για τον προπολογισμό τη κοινωνική Ευρώπη. Χρησιμοποιήστε τα λοιπόν όλα αυτά. Αξιοποιήστε αυτέ τι ιδέε. Σα ευχαριστώ και να με συγχωρείτε που μακρηγόρησα. Ναι. Η πρόεδρο, να μου επιτρέψετε να ε, αναγνώσω τα ονόματα από την λίστα για τα πρόσωπα που επιθυμούν να ερωτήσουν. Θα ακούσουμε τώρα δηλαδή την κυρία Οραν Σατσί, μετά ο κύριος Σούλτσε και μετά η κυρία Αρένα. Όμως πρώτα θα δώσω τον λόγο στον Υπουργό για να μπορέσει να απαντήσει τις ερωτήσεις Πυρίνσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με όσα εξήγησε ο κ. Πύρινς. Όντως διανύουμε μια ε, περίοδο βελτίωση των οικονομικών και αυτό θα πρέπει να το αισθανθούν όλοι. Ωστόσο, ο ευρωπαϊκός πυλώνας, ο ευρωπαϊκός κοινωνικός πυλώνας ήταν κάτι καλοδεχόμενο λοιπόν από την άποψη αυτή. Όπως είπα, πέρσι τον Νοέμβριο υπογράφτηκε διακήρυξη στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας. Ήρθε η ώρα τώρα να εφαρμοστούν οι προβλέψεις εκείνης της διακήρυξης, να γίνει προσπάθεια δηλαδή να υλοποιηθούν και αυτό είναι μία από τις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας. Ε, σχεδιάζουμε να εμφυσίσουμε πνοή ε, σε αυτό το σχέδιο ήδη από την πρώτη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σε ένα από τα σημαντικότερα διαβήματα που θα κάνουμε μέσα στην Προεδρία μας έχουμε και τον σχεδιασμό για να οργανώσουμε μια ε, διάσκεψη για νέα ευρωπαϊκά πρότυπα στον ε, κοινωνικό τομέα. Θα επανεξετάσουμε τα όσα έχουμε ήδη σε ό,τι αφορά τον ε, Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και βέβαια αυτό θα τεθεί στη συζήτηση και στην τριμερή διάσκεψη του Μαρτίου θα θέσουμε δηλαδή και εκεί το θέμα αυτό. θα εντάξουμε τον κοινωνικό πυλώνα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, αυτό είναι το ένα θέμα. Και δεύτερο, θα επανεξετάσουμε τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και μέσα στα πλαίσια του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου, κάτι που θα μας επιτρέψει να προβλέψουμε μια χρηματοδότηση για την επόμενη ε, χρηματοδοτική περίοδο υπέρ της κοινωνικής Ευρώπης. Τώρα για την άλλη σας ερώτηση, δηλαδή την εγγύηση υπέρ των παιδιών. Αυτό και για μας είναι πολύ σημαντικό θέμα. Πρόκειται για πολιτική συζήτηση που είναι σημαντική ε, από μόνη της, δεν είναι δηλαδή μονάχα ο μηχανισμός χρηματοδότησης. Ε, είπα ήδη ότι η ανάπτυξη της παιδικής ηλικία, η εξέλιξη της παιδικής ηλικία δηλαδή, είναι πολύ σημαντική ήδη και εκεί θα προβλέψουμε και επένδυση, επενδύσεις δηλαδή, χρηματοδότηση. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό η παιδική ηλικία για όλες και όλους. Συμφωνώ άλλωστε μαζί σας ότι η μελλοντική Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα παίξει σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει να μπορέσει να βασιστεί στα μέχρι τώρα επιτεύγματα μεταξύ αυτών, αυτών δε και το έργο που έχει κάνει η πλατφόρμα για την αδήλωτη εργασία. Θα είναι σημαντική και η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Εκεί επίσης θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε με επιτυχία το έργο, επιτυγχάνοντας συνένεση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Τώρα για την οδηγία, για την εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή, που και αυτό αποτελεί προτεραιότητα της ε, Βουλγαρικής Προεδρίας, εκεί έχω να πω ότι το έργο, ή μάλλον η εργασία για το θέμα αυτό είναι ήδη πολύ σημαντική και για την υλοποίηση του κοινωνικού πυλώνα. Οι δε προσπάθειές μας θα στοχεύσουν στο να επιτευχθεί μια συνολική προσέγγιση από πλευρά Συμβουλίου ήδη βεβαίω από την επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Υπουργών. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε, κύριε Υπουργέ. Η κυρία Μωράν Σαρτιέ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Είμαι εισηγήτρια για την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων και οφείλω να σας πω ότι αναλαμβάνετε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έλεγα με θάρρος. Έχουμε δικαίωμα από την αρχή της Προεδρίας σας να χαρούμε την ε, επίσκεψη του Πρωθυπουργού σας κ. Μπορισόφ. Είστε και εσείς ε, σήμερα εδώ μπροστά μας. Η Υφυπουργός σας κ. Μπρουσίνοβα ήδη ε, συνεργάζεται μαζί μας και κάποιος είπε ότι ήταν και στον τριμερή διάλογο αλλά δεν ήταν ε, που είμαστε μαζί με την κυρία Γιονγκέριους μπορούμε να σα πούμε τα σχετικά και θα σα πούμε και τι σκεπτόμαστε σχετικά. Θεωρώ ότι έχετε μεθοδικότητα στην εργασία σας, έχετε επαγγελματισμό στις διαπραγματεύσεις, ιδίως έχετε όμως ανοιχτό πνεύμα που μπορεί να μας επιτρέψει να προχωρήσουμε για ένα θεμελιώδε κείμενο όπως αυτό της οδηγίας απόσπαση εργαζομένων που μας απασχολεί και επί του οποίου επιθυμούμε απολύτω να επιτύχουμε ε, μια σημαντική καμπή ε, στην Ευρώπη που είναι βεβαίως ε, σχετική και με τον κοινωνικό πυλώνα. Αυτό ακριβώς κάνουμε ως κοινή προσπάθεια με την επεξεργασία της εν λόγω οδηγίας και οφείλω να πω ότι για μένα δεν υπάρχουν μικρές και μεγάλες χώρες. Όταν βλέπω μια χώρα όπως η Βουλγαρία που εμφανίζεται όχι ως Βουλγαρία αλλά ως πραγματική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πραγματική βούληση να συμμετάσχει στην οικοδόμηση της Ευρώπης εγώ σας λέω συγχαρητήρια και είμαστε διατεθειμένες να ε, βαδίσουμε μαζί σας στην κατεύθυνση του οράματος αυτού, όπως είπε προηγουμένως και η συνάδελφός μου Τζιν Λάμπερτ, μικρή δυναμική χώρα. Υπάρχουν και άλλες χώρες μεγάλες, θεωρούν ότι είναι μεγάλες, αλλά δεν έχουν την ίδια βούληση ε, να εργαστούν. Θα ήθελα να θέσω τώρα τρία θέματα. Το πρώτο είναι πράγματι, επανέρχομαι, η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Ζήτημα όπου θα πρέπει να συμπαραταχθεί η Ευρώπη ε, με τις δικές μας προσπάθειες. Έτσι, με αυτό το πνεύμα κινούμεθα, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δύσκολο στο Συμβουλίο, βεβαίως και στο Κοινοβούλιο ήταν περίπλοκα τα πράγματα. Είμαστε, όσοι γνωρίζετε, 751 ευρωβουλευτές από 8 διαφορετικές κοινοβουλευτικές ε, παρατάξεις και βεβαίως ε, θέλουμε διάλογο μαζί σας, διαβούλευση και μέσα από αυτά έχουμε επιτύχει διαπραγματευτική, ε, διαπραγματευτική εντολή ε, ισχυρή. Τώρα, οι ομάδες που εργάζονται στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την κυρία Γιονγκέριους, η κυρία Τάισεν από την Επιτροπή και η Υφυπουργός σας κυρία Ρωσίνοβα. Όλη αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να γίνει για να ε, οικοδομήσουμε και μια συμφωνία, αλλά θα χρειαστεί επίση και θα πρέπει να το υποσχεθούμε αυτό, ότι ε, θα ρίξετε το βάρος σας στις προσπάθειες ώστε να ε, επίστε το Συμβούλιο να συνεργαστεί. Όλοι αυτοί οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που άλλα λένε στις χώρες τους και άλλες θέσεις λαμβάνουν στο Συμβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν να δείξετε πραγματική ηγετική ικανότητα απέναντι σε όλες τις χώρες που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο και θα πρέπει να τους συμπαρασύρετε ας πούμε όλους αυτούς. Αυτή είναι η εκκλησή μου διότι στα χέρια σας βρίσκεται εν μέρη η επιτυχία της προσπάθειάς μας. Και εμείς οι συνεισηγήτριες θα σας υποστηρίξουμε. Αλλά και εσείς πρέπει να κάνετε το δικό σας καθήκον στο Συμβούλιο. Δεύτερον, Ε, ε, Βεβαίω μια καμπή στην απασχόληση. Είπατε ότι η απασχόληση είναι μια, ένα από τα θέματα που σα απασχολούν. Βεβαίω όλε και όλου μας. Όμως σήμερα η εξέλιξη τη της απασχόλησης της των αναγκών, των, ε, γενικώ εξέλιξης της απασχόλησης έχει ανάγκη από βαθιές αλλαγές ό,τι αφορά κυρίως την εκπαίδευση. Η αρχική εκπαίδευση ε, δεν αρκεί πλέον για να καλύψει ανάγκες ανάγκε των επιχειρήσεων. Πρέπει να επιταχύνομαι. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο ρωτώ αν πρόκειται να προωθήσετε μια νέα πολιτική για την εξέλιξη, την ανάπτυξη των ε, επαγγελματικών δεξιοτήτων που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις και ε, μάλιστα δεξιότητες που να μπορούν να μεταφέρει ο εργαζόμενος και αλλού. Το τρίτο, άλλο μέγα κοινωνικό θέμα που είναι η εξορρόπηση της ε, ε, επαγγελματικής με την προσωπική ζωή. Και σε αυτό το κείμενο θα πρέπει να εγγύψετε με πολύ σοβαρό τρόπο, διότι μιλούμε για την ισότητα στην εξέλιξη των σταδιοδρομιών. Στην ισορροπία επαγγελματικού και προσωπικού βίου θα πρέπει εσείς να εγγύψετε στις επιπτώσεις αυτής της υφιστάμενης έλλειψης ισορροπίας στις σταδιοδρομίες των γυναικών. 61% των πτυχιούχων στο ευρωπαϊκό επίπεδο σήμερα είναι γυναίκες. Άρα υπάρχει μια πλειοψηφία πτυχιούχων γυναικών. Αν όμως εξετάσετε τις σταδιοδρομίες τους, υστερούν απέναντι σε αυτές των ανδρών. Σας ευχαριστώ λοιπόν εξ ονοματοστόλων των γυναικών που θα ε, στρέψετε την πολιτική σας προσπάθεια γύρω από την λήψη υπόψη αυτής τη ε, ανισορροπία. Και βεβαίω, αν τα πράξετε όλα αυτά θα έχετε κερδίσει την εμπιστοσύνη μας. Thank you, ε, Mr. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργό, κύριε Πέτκο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την απόσπαση των εργαζομένων για όσα είπε. Είναι ένα θέμα που απαιτεί δύσκολες διαπραγματεύσεις. Εγώ συμμετείχα στους δύσκολους συμβιβασμούς που πετύχαμε τον Οκτώβριο στο Λουξεμβούργο και ξέρω πόσο δύσκολο ήταν να καταλήξουμε σε αυτό το συμβασμό. Ξέρω πόσες ελπίδες είχαν βάλει όλες οι πλευρές αυτό το θέμα. Πάντως έχει μεγάλη σημασία. Μεγάλη σημασία έχει η κοινωνική προστασία των αποσπασμένων εργαζόμενων, αλλά και η διατήρηση της ελευθερίας προσφοράς υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παροχής υπηρεσιών. Καμία αμφιβολία δεν υπάρχει. Για να πετύχει κανείς σίγουρα χρειάζεται ηγεσία. Και δεν νομίζω ότι αυτό θα λείψει στην ομάδα της Βουλγαρικής Προεδρίας που θα δουλέψει πάνω σε αυτό το θέμα. Σας είπα ποιες είναι οι προτεραιότητές μας και μία από αυτές είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτεί η σημερινή αλλά και η αυριανή αγορά εργασίας δεξιότητες που να μεταφέρονται επίσης από τη μία χώρα στην άλλη. Πολλές φορές έχω υπογραμμίσει πόσο μεγάλη σημασία έχει και η οδηγία η οποία προσπαθεί να πετύχει ισορροπία ανάμεσα στην ε, προσωπική και την επαγγελματική ζωή. Είναι ένα καλό παράδειγμα ε, η προσπάθεια αυτή να πετύχουμε ισορροπία και ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Βουλγαρία είναι μια χώρα που σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές το ποσοστό των εργαζόμενων γυναικών στις τεχνολογίες επικοινωνιών είναι το υψηλότερο από οπουδήποτε αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την Eurostat. 27 100 των γυναικών δουλεύουν σε αυτό το κλάδο, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 16%. Και αυτό είναι πολύ βασικό για μας. Αυτό μπορώ να πω λοιπόν για να απαντήσω την ερώτησή σας για αυτό που έθεσαν οι αξιότιμοι ευρωβουλευτές σας. Πρόεδρος, παρακαλώ. Τώρα εσείς. Κύριε Σούλτσε. Κύριε Υπουργέ και εσείς κυρία Υφυπουργέ, σας ευχαριστώ για την ελευσή σας σήμερα εδώ. Καλό μάλιστα είναι που έρχεστε ως δίδυμο και ε, ε, είμαι Γερμανός ε, και νομίζω ότι ε, είναι ανεξάρτητο το αν προέρχεται κανεί από μεγάλη ή μικρή χώρα. Το ζήτημα είναι αν θα κάνει μια καλή ή όχι καλή προεδρία. Τα τελευταία χρόνια είδαμε στην Ευρώπη κατ' επανάληψη μικρέ χώρε να ασκούν πολύ καλά την προεδρία. Είδαμε όμω και άλλε, και δεν εννοώ την Εστονία, εννοώ άλλη προηγούμενα από αυτήν που δεν τα κατάφερε και τόσο σπουδαία. Σήμερα εσείς ε, αναπτύξατε πολλούς στόχους που επιθυμείτε να επιτύχετε μέσα σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ε, των έξι μηνών. Είμαι όμως πεπισμένος ότι επειδή αναλαμβάνετε για πρώτη φορά την Προεδρία από την ένταξή σας, θα εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία αυτή. Δύο θέματα θέλω να σας ε, θέσω. Αφενός τον κανονισμό 883, συντονισμό των κοινωνικών συστημάτων είπατε ότι το ζήτημα των ε, ε, επιδομάτων ανεργίας και άλλων στήριξεων για την ανεργία θα είναι πολύ σημαντικό για την Προεδρία σας. Ποια είναι τώρα και η θέση σας σχετικά με τη μετατροπή, με την, ε, με την αλλαγή έδρας και την μεταφορά των δικαιωμάτων για την ανεργία. Το άλλο θέμα είναι η διασύνδεση με τον τιμάριθμο των ε, επιδομάτων τέκνων. Στην έκθεσή της δεν το έχει περιλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιζητούμε συζήτηση. Έχουμε την κατάσταση τώρα ότι ανάμεσα σε μεγάλες σημαντικές, ασφαλώς είναι όλες οι, Ευρω... όλες οι χώρες μέλη της Ένωσης σημαντικές, υπάρχουν όμως χώρες όπως Αυστρία, στην Γερμανία διεξάγεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των, των επιδομάτων τέκνων. Δεν γνωρίζω ποια είναι η στάση της Βουλγαρίας προκειμένου, αλλά πώς θα αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό τους επόμενους μήνες. Δεν μπορεί κανείς απλώς να πει το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Έχουμε μια κατάσταση πολύ περίπλοκη και ευαίσθητη. Έχουμε διάσταση απόψεων ανάμεσα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ερώτημά μου είναι πώς θα διαμεσολαβήσετε εν ώψη και του γεγονότος ότι ε, ο διάδοχός σας στην ε, Προεδρία του Συμβουλίου θα είναι η Αυστρία. Ε, με ενδιαφέρει λοιπόν πολύ το πώς αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας για τον κανονισμό αυτών. Το σύστημα συντονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα δουλέψουμε σκληρά προκειμένου να πετύχουμε μια κοινή προσέγγιση στο Συμβούλιο. Και μια στο μερική κοινή προσέγγιση στα υπόλοιπα κεφάλαια του κανονισμού για το επίδομα ανεργίας για παράδειγμα όπου υπάρχουν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχουν να κάνουν με την μεταφορά τέτοιων ε, επιδομάτων μεταξύ χωρών. Από τη χώρα που το οφείλει προς την χώρα που κατοικεί ο δικαιούχος. Είναι μια συζήτηση παραμένει ανοιχτή στο Συμβούλιο. Θα συζητήσουμε με κάθε λεπτομέρεια τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το κεφάλαιο του κανονισμού. Όσον αφορά τώρα τα οικογενειακά επιδόματα, συζητήθηκαν το Δεκέμβριο στο Συμβούλιο. Και εκεί υπήρξε συμφωνία για μια μερικώς νέα προσέγγιση. Το θέμα της τιμαριθμικής προσαρμογής δεν τέθηκε προς το παρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θα το θέσουμε ούτε εμείς, δεν σκοπεύουμε. για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή και το συντονισμό τους. Πάντως, τονίζω ξανά και ξανά ότι κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας και εν ώψη των ευρωεκλογών που μετά θα έχουμε νέο κοινοβούλιο και νέα επιτροπή να ξέρετε ότι στο μεταξύ θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτευχθεί συμφωνία πάνω σε αυτήν την τόσο σοβαρή υπόθεση που είναι ο συντονισμός των κοινωνικών συστημάτων στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Η Μαρία Ρένα έχει την τελευταία ερώτηση, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ. Εκτίμησα πολύ τόσα μας είπατε και τις διάφορες πρωτοβουλίες, είτε την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων, είτε για την ε, συμφιλίωση της προσωπικής με την επαγγελματική ζωή. Νομίζω ότι η Βουλγαρική Προεδρία μπορεί να περάσει από το σλόγγαν που λέει «Χάνουμε τη ζωή μας για να την κερδίσουμε», τελικά κερδίζουμε τη ζωή μας για να τη ζήσουμε καλύτερα. Ελπίζω τουλάχιστον αυτό να πετύχουμε, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ναι, να κερδίσουμε τη ζωή μα δουλεύοντα, αλλά για να τη ζήσουμε καλύτερα. Να τη ζήσουμε καλύτερα όταν είμαστε αποσπασμένο, όπου έχουμε την εντύπωση ότι σε αυτή την υπόθεση αντιπαραθέτουμε τις χώρες της Ανατολής και της Δύσης, τις χώρες του Βορρά και του Νότου, μα όποιος και να είναι ο εργαζόμενος, στόχος μας πρέπει να είναι να τον προστατεύουμε, να μπορεί να συνεχίσει να κερδίζει τη ζωή του, αλλά να την κερδίζει για να μπορεί να τη ζήσει καλά. Και αν η Βουλγαρική Προεδρία μπορεί να εγγραφεί σε αυτή τη λογική, νομίζω ότι όλοι θα έχουμε να κερδίσουμε, όποια και αν είναι η πολιτική άποψη του καθενός. Το δεύτερο ζήτημα που έχει να κάνει ακριβώς με αυτό, με το πώς θα κερδίσουμε τη ζωή μας για να τη ζήσουμε καλύτερα, είναι ο συνδυασμό της οικογενειακής και της επαγγελματική ζωής. Πάνω από 55% των εργαζομένων σήμερα δύσκολα μπορούν να διαχειριστούν την προσωπική του ζωή με την επαγγελματική. Διαπιστώνουμε πάρα πολλές περιπτώσεις burnout στις επιχειρήσεις διαπιστώνουμε ότι πτωχεύει η κοινωνική ζωή των εργαζομένων γιατί τελικά δεν τους μένει χρόνος να κάνουν τίποτα άλλο από το να δουλεύουν. Οπότε η οδηγία αυτή πρέπει οπωσδήποτε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες αυτού του 55% των εργαζομένων. Και αν το καταφέρουμε, τότε ανταποκρινόμαστε και στις επιθυμίες των επιχειρήσεων. Γιατί οι επιχειρήσεις τι είναι, αν δεν έχουν τους μισούς τους εργαζόμενους δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει με το από ποια οικογένεια πολιτική ερχόμαστε ή κόμμα. Όχι, όπως στηρίζουμε τους εργαζομένους, στηρίζοντας άρα τις επιχειρήσεις, γιατί είναι τα αυτά τα δύο. Και αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε και ελπίζουμε να το πετύχετε και εσείς στο Συμβούλιο. Και το τρίτο το θίξατε, αλλά κάπω ιδιαίτερα. Είναι το θέμα της απασχόλησης σε συνδυασμό με την ψηφιακή οικονομία. Πρέπει να δούμε πώς οι γυναίκες μπορούν να εκπροσωπηθούν καλύτερα στην ψηφιακή οικονομία. Αυτό που εμένα με απασχολεί στην ψηφιακή οικονομία είναι περισσότερο το θέμα του καθεστώτος. Και εδώ διαπιστώνουμε ότι έχουμε όλο και περισσότερους νέους εργαζόμενους οι οποίοι ε, σκοτώνονται στη δουλειά χωρίς ειδικό καθεστώς, χωρίς κοινωνική προστασία, χωρίς δικαιώματα. Οπότε εδώ πρέπει η Ευρώπη να αποδειχτεί σύγχρονη. Δεν είναι δυνατόν να βάζει τους εργαζόμενους αυτούς σε μια μορφή σκλαβιάς όπως είχαμε στο 19ο αιώνα. Όχι, πρέπει και εδώ να προστατεύσουμε και αυτούς τους εργαζόμενους της ψηφιακής οικονομίας. Οπότε για αυτές τις τρεις υποθέσεις είπατε τι θέλετε να κάνετε, αλλά ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά σας προκειμένου τελικά το Συμβούλιο να πάψει να συμπεριφέρεται με τέτοια ε, συστολή, αλλά να μπορέσει να ανακτήσει ο κόσμος την εμπιστοσύνη του σε αυτά που γίνονται από την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση για τώρα. Σωρή ερωτήσεων θα έχετε το επόμενο εξάμεινο. Αλλά για την ώρα αυτή είναι η τελευταία. Κύριε Πέτκοφ. Ευχαριστώ κυρία Κόκ. Οπωσδήποτε. Οι ερωτήσεις που μόλις ακούσαμε είναι πολύ σημαντικές γιατί αφορούν τους εργαζόμενους. Στα πλαίσια της ψηφιακής οικονομίας αγείρονται σημαντικά ζητήματα. Να τονίσω ότι μια από τις βασικές προκλήσεις που θα έχει να αντιμετωπίσει η αγορά εργασία στην Ευρώπη θα είναι ακριβώ ο εξυγχρονισμός των συμβάσεων εργασίας και των ε, σχέσεων μεταξύ εργοδότη εργαζομένου. Πρέπει να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή διαλεκτικότητα για τις εταιρείες αλλά να διαφυλάξουμε τις καλές εργασιακές συνθήκες εντός αυτού του χώρου. Ένας τρόπος να το πετύχουμε αυτό θα είναι η οδηγία για τις ε, διαφανείς και προβλέψιμες εργασιακές συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προτάθηκε πέρσι. Η οδηγία αυτή θα μας βοηθήσει να πετύχουμε μερικούς από τους στόχους μας στο επίπεδο του κοινωνικού πυλώνα. Στόχους που έχουν να κάνουν με την ε, ευελιξία και τις ευέλικτες εργασιακές συνθήκες, καθώς και την προστασία σε περιπτώσεις απόλυσης. Η πρόταση αυτή οδηγίας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων της Βουλγαρικής Προεδρίας. Επιπλέον, ήδη ανέφερα προηγουμένως ότι η εξισορρόπηση επαγγελματικού ιδιωτικού βίου είναι από τις βασικές προτεραιότητες που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προχωρήσουμε. Όσο πιο πολύ μπορούμε. βλέπουμε πώς θα φροντίσουμε τα μέλη της οικογένειας, τι κάνουμε με τους φροντιστές άλλων μελών της οικογένειας και τι γίνεται με όσους ταξιδεύουν, πώς μπορούν να συνδυάσουν τις επαγγελματικές και τις προσωπικές τους υποχρεώσεις. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας ιδιαίτερα γιατί είναι πολλές οι χώρες όπου οι γονεί αναγκαστικά απουσιάζουν από την εργασία. Η τιμωρία του είναι να φροντίσουν τα παιδιά του. Και αυτό είναι ένα πλήγμα για την αγορά εργασία. Υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Η εξισορρόπηση λοιπόν επαγγελματικού ιδιωτικού βίου είναι άκρο σημαντική για την ε, ευρωστία της αγοράς εργασίας. Και αυτό σε σχέση με τις δημογραφικές απειλές που αντιμετωπίζουμε και τις απαιτήσει στην αγορά εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας και σας ευχαριστούμε για το θερμό καλωσόρισμα στην Επιτροπή σας σήμερα. And Η Πρόεδρος Ουλσκόπ, σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την σημερινή παρουσία σας εδώ και επίσης σας ευχαριστώ για το γεγονός που μας δώσατε πραγματικές απαντήσεις στις ερωτήσεις. Ναι. Ε, σας ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι και ευχαρίστως θα σας ξαναδούμε. Θα σας ξαναέχουμε κοντά μας. Thank a question. Uh,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 Okay, friends. Η πρόεδρος. Δεν έχουμε ακόμη τελειώσει. Ακολουθεί το επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης, το οποίο είναι το υπαριθμονικό 23, κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχολήσεις των χωρών μελών. Πρόκειται για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και για το θέμα αυτό εννοώ. Και εάν υποσχεθείτε ότι δεν θα κάνετε προσωπικούς διαλόγους χωρίς ε, να σας δώσω το λόγο βέβαια πρώτα, θα δώσω τον λόγο πρώτα στην κυρία Σντάνοκα, η συγγήτρια. Ορίστε κυρία Σντάνοκα, έχετε το λόγο, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, Όλοι νομίζω εντυπωσιαστήκαμε από την ανταλλαγή απόψεων με τον εκπρόσωπο της Προεδρίας. Ακούσαμε βέβαια και πολλές ευχές. Ελπίζω και το θέμα το, το οποίο φέρω την ευθύνη εγώ να δηλαδή για την επεξεργασία του να μην ελπίζω να ληφθεί υπόψη σοβαρά από το Συμβούλιο. Το θέμα εδώ είναι δυστυχώς η έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου, διότι εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απλώς ακούεται, δηλαδή δεν έχει πλήρη εμπλοκή. Ελπίζω να μην έχουμε μια κατάσταση όπως τα προηγούμενα χρόνια όπου τα σχόλιά μας σχεδόν δεν λαμβάνονταν καθόλου υπόψη. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να συντάξουμε ένα κείμενο με κοινή προσπάθεια με μεγάλη στήριξη από την Επιτροπή Απασχολήσεως να ακουστεί δηλαδή δυνατή η φωνή μας απέναντι στο Συμβούλιο, το οποίο βεβαίως θα χρειαστεί και να την ακούσει και να την προσέξει. Γι' αυτό θα ήθελα πρώτα να ακούσω προσεκτικά τα σχόλια των ε, σκιωδών εισηγητών και έτσι να μπορέσω να συντάξω το έγγραφο για την περαιτέρω συζήτηση. Πρώτη λοιπόν αποτίμηση της ε, προτάσεως της Κομισιόν είναι θετική. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Αποδίδεται μεγαλύτερη έμφαση στα κοινωνικά δικαιώματα, στις ίσες ευκαιρίες, στην κοινωνική προστασία και συμπερίληψη, το δικαίωμα να έχει κανείς κάποιο ελάχιστο εισόδημα. Αυτές είναι οι ιδέες τις οποίες υποστηρίζει εδώ και πολύ καιρό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. προβλέπεται και η διασύνδεση με τον κοινωνικό πυλώνα. Σωστό. Αυτό θα πρέπει να γίνει όμως μέσα σε όλο τον κύκλο των ειδικών συστάσεων αναχώρα. Σωστό είναι που υπάρχουν και νέοι κοινωνικοί δείκτες και το λεγόμενο βαθμολόγιο όμως δεν είναι επαρκής διότι δεν καλύπτουν όλες τις πτυχές του ευρωπαϊκού κοινωνικού πυλώνα ούτε έχουν επαρκή δύναμη για να επιφέρουν τις αναγκαίες διορθώσεις. Είμαστε αποφασισμένες να περιλάβουμε στο κείμενο με σαφέστερο τρόπο την ανάγκη να αντιμετωπιστεί ο κοινωνικός αποκλεισμός καθώς και όλες οι μορφές φτώχειας, να αναπτύξουμε τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις που ιδρύουν μετανάστες, να δημιουργήσουμε μια ε, ενιαία αγορά πιο ισορροπημένη και χωρίς αποκλεισμούς, με επαρκή κοινωνική προστασία και τέλος να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην απασχόληση. Αυτά που είπα τώρα είναι η βασική μας στόχοι που θα περιληφθούν στο κείμενό μας. Λοιπόν, θα αρκεστώ σε αυτά και αναμένω να ακούσω τα σχόλια των εκπροσώπων των άλλων πολιτικών ομάδων. Η Πρόεδρος Ούλουφ Σκόμπ Θα δώσω το λόγο στο νέο μέλος της Επιτροπής μας, Μικαήλ Ντέτσιν, που αντικαθιστά την Ιούτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Συγήτρια για την παρουσίαση του θέματος. Ευχαριστώ, θα συνεργαστώ μαζί σας. Για μένα δύο πράγματα είναι σημαντικά. Πρώτα, η πρόταση του Συμβουλίου αναφέρεται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα Δικαιωμάτων. Σωστή αφετηρία αυτή. Αυτό που βρίσκω να λείπει είναι η εξίσωση των οικονομικών με τα κοινωνικά δικαιώματα όλων των πολιτών κοινωνικά δικαιώματα, κοινωνικά συμφέροντα δεν θα πρέπει να αντιπαρατάσσονται στα οικονομικά. Αυτό είναι νομίζω σημαντικό. Οι κοινωνικοί δείκτες στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, καθώς και οι ειδικέ αναχώρα συστάσεις, θα πρέπει να αναδειχθούν εντονότερα. Να κάνουμε και προτάσεις για τις χώρες μέλη δηλαδή. Συμφωνώ με την προλαλή σας απάντως. Από το 2015 δεν υπάρχουν τροποποίησεις στην πολιτική απασχόληση και στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές. Χαίρομαι πάντως που το Συμβούλιο φαίνεται να ακολουθεί τις υποδείξεις του Κοινοβουλίου και ιδίως σε ό,τι αφορά την θέσπιση κατώτατου εισοδήματος. Αποδέχεται την αξίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Συμβούλιο. Αυτό είναι θετικό σημάδι από την πλευρά του Συμβουλίου. Και σε ό,τι αφορά τις κατευθείας γραμμέ της πολιτικής απασχόλησης, θα απευθύνω και εγώ έκπληση προς το Συμβούλιο να μην αγνοήσει τούτη φορά τα όσα λέει το Κοινοβούλιο η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Δεν έδωσα τον λόγο στον Μάρεκ Πλούρα, αλλά φαίνεται πως δεν τον αντικαθιστά κανείς και είναι απόν. Θα ακολουθήσει η κυρία Τρεμπέσιους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι κατευθυντήρες γραμμές για μέτρα πολιτικής της απασχόλησης των χωρών μελών 2017 δεν είναι βεβαίως και η πρώτη έκθεση του είδους αυτού. Απέναντι σε προηγούμενες εκθέσεις, εδώ αυτό που διαπιστώνω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υποτίθεται ότι θα αναλάβει μεγαλύτερε ευθύνε. Στην παράγραφο 2 μιλούν για το αμφισβητούμενο θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού, την ισότητα των δύο φύλων και από αυτό απορρέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναμειχθεί σε πολλά θέματα της απασχόλησης όπως για παράδειγμα εγγύηση μιας πρέπουσας κοινωνικής εγγύησης. Δηλαδή αυτό το ελάχιστο εισόδημα του Χάρτς 4 στην Γερμανία. Πώς είναι δυνατόν να προσπαθούν να επανέρχονται διαρκώς σε κάποιες, στην προώθηση κάποιων σοσιαλιστικών μοντέλων Προ τα κάτω εξίσωση. Θα έπρεπε να είχαμε διδαχθεί κάτι από την ιστορία μα. Και αυτό που βλέπουμε ωστόσο είναι τα ίδια και τα ίδια. Μακάνε μου τέτοια πράγματα. Πολιτική τη απασχόληση και πολιτική κοινωνική θα πρέπει να παραμείνουν στην αρμοδιότητα των χωρών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπεται να αναλάβει εγγυήσει για κοινωνική στήριξη. Και αν το πράξει αυτό, τότε πρώτα να απαντήσει στο ποιο θα καλύψει το κόστο. Δεν θέλουμε το θέμα του κόστους να αχθεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι υποθέσει των χωρών μελών και αυτές θα πρέπει να λυθούν μέσα στα πλαίσια της επικουρικότητας. Μιλούν επίσης για κρατικές δαπάνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προτείνει δαπάνες των κρατών μελών. Οι χώρες μέλη και ιδίω τα μέλη της Ευρωζώνης θα πρέπει πρώτα να φροντίσουν να εξηγιάνουν τους προϋπολογισμούς τους. Εάν έχουν κάποια περιθώρια, α τα χρησιμοποιήσουν στου δύσκολου καιρού. Εάν δεν υπάρχει δημοσιονομική πειθαρχία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προτείνει αντικυκλικές δαπάνε και ιδίω όχι όταν αυτά οδηγούν ξανά και ξανά στην παραβίαση των κριτηρίων για τα ελλείμματα. Πολλοί μιλούν για αύξηση των ευθυνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά όμως είναι σαφής προσπάθεια παραβίασης της αρχής της επικουρικότητας. Αναμένω το κείμενο της εισηγήτριας, το οποίο ε, ωστόσο εγώ θα ταχθώ απέναντι πάρα πολύ επικριτικά. Ευχαριστώ. Άννα Τούμ δεν είναι παρούσα, δηλαδή μπορούμε να προχωρήσουμε. Α, εσείς την αντικαθιστάτε, κύριε Σαμπόν, μάλιστα. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. όντω την αντικαθιστώ εγώ, θα είμαι σύντομο. Τώρα βέβαια μιλάω μετά από την κυρία Τρουπέσιους, ίσως αν είχε μιλήσει μετά από μένα να μην είχε αντιταχθεί σε αυτά που λέω, αλλά πάση περιπτώσει πολύ απλά λέω ότι εγώ θέλω να πω τα αντίθετα από αυτά που είπε εκείνη. Εγώ πιστεύω στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, εγώ πιστεύω στο ευρωπαϊκό μοντέλο, εγώ πιστεύω ότι πρέπει οπωσδήποτε να καθορίσουμε ένα level playing field, δηλαδή οι ισότιμες συνθήκες για τον ανταγωνισμό, τον θεμητό ανταγωνισμό, έτσι, να παίζουμε ένα παιχνίδι ομοιογενές και όχι με άνισες ευκαιρίες. Αλλιώς η Ευρώπη θα σπάσει, δεν θα αντέξει. Βέβαια, εύχομαι πολύ κουράγιο στην εισηγήτρια και θα ολοκληρώσω με το εξή. Όπως οποιοδήποτε άλλο έγγραφο γενικής φύσεως, στρατηγικής που έχει να κάνει με την απασχόληση, είναι προφανές ότι πρέπει να προσανατολιστεί στην εφαρμογή στην πράξη των όσων συμφωνήθηκαν στο Γκέντανμπουργκ. Δηλαδή, κοινωνικός πυλώνας της Ευρώπης. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πάμε. Έχουμε ένα μοντέλο, έχουμε μια επιθυμία, έμπνευση, τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμά. Οπότε, τώρα, με κάθε δυνατό τρόπο, πρέπει να φροντίσουμε, είναι χρέος μας, σιγά σιγά να τα εφαρμόσουμε και στην πράξη. Και αυτά ζητάω από την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο Πατρίκ δεν είναι εδώ. Κάποιος άλλος από την ΚΟΕΠ πως τον αντικαθιστά. Όχι. Ωραία. Η FDD τώρα, η Λαράκας δεν είναι εδώ, ούτε την αντικαθιστά κανείς από ό,τι βλέπω. Η ΕΝΕΦ. Ο κύριος Μαρτάν. παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι έχει πολύ θάρρος η συγκήτρια που ασχολείται με ένα τέτοιο θέμα που επανέρχεται συνέχεια για τις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την απασχόληση, κατευθυντήριες γραμμές προς τις χώρες μέλη. Και νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια υπερβολή. Καταλαβαίνω, ο κύριος Καλβεσαμπών μας είπε πω τι ευκαιρία είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. ναι, αλλά τελικά ε, ανάλογα με το πώς ξεκινάνε φτιάχνει το τοίχο, ε, κρίνουμε το πόσο καλό είναι ο χτίστης. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα, κύριε Καλβέ. Πλήρης απασχόληση, η απόφαση του Συμβουλίου Πολέμηση της ανεργίας του κοινωνικού αποκλεισμού, δεύτερο. Ναι, ωραία, κύριε Καλβέ Σαμπό και κυρία Συγήτρια. Εντάξει, οι στόχοι μπορεί να είναι απόλυτα θεμητοί. Ποιο δεν θέλει να καταργήσει την ανεργία. Ποιο δεν θέλει να βελτιώσει τη λειτουργία των αγορών ε, εργασία, Ποιο δεν θέλει να αναπτύξει τον κοινωνικό διάλογο, όπω λέει τη γραμμή 7, ή να ευνοήσει την κοινωνική ένταξη και να καταπολεμήσει τη φτώχεια, όπως προτείνει η κατευθυντήρια γραμμή 8. Ποιος δεν τα θέλει όλα αυτά. Αλλά κύριε Συγγήτρια, καταλαβαίνω ότι είσαστε απογοητευμένοι διότι αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για ένα κατάλογο ευσεβών πόθων. Πρόκειται για ένα κατάλογο όπου μαζί με τον κύριο Γαλβέ Σαμπόν όλοι στην ουσία είμαστε υπέρ. Με έξι ίσως θα μπορούσαμε να τα είχαμε καταφέρει, αλλά έτσι όπως φουσκώσαμε και γίναμε 28 Συνοχή, πού να τη βρούμε. 28 είμαστε ακόμα, τι να κάνουμε. Σύγκληση, πούντα. Κατεβαίνουμε, ισοπαίδωση προς τα κάτω. Τι μέσα έχουμε για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, ανάπτυξη της ενίας αγοράς, περισσότερη κινητικότητα, ε, κανένας οικονομικός πατριωτισμός, ε, μεταρρυθμίσεις διαφθρωτικές... βάση της κατευθυντής γραμμής 6 με τρελιτότητα σας υπενθυμίζω, ή ακόμα και επιδοτήσεις, ξέρω ότι σας ενοχλεί, που δίνονται στους πρόσφυγες, όπως το εξηγεί το σημείο 3.1 της στρατηγικής που περιλαμβάνει η έκθεση Επιτροπής και του Συμβουλίου, που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ετήσια εξέταση της ανάπτυξης 2018. Αυτά είναι που εμείς καταγγέλουμε. Αυτά είναι που διαπιστώνετε κι εσείς. Η έκθεση αυτή εξάλλου αντιφάσκει. Γιατί, κυρία Συγκίτρια, λέει ότι οι κοινωνικές δυσκολίες έχουν την τάση να μεταφέρονται από τη μία γενιά στην επόμενη. Και ο κίνδυνος αυτός, λέει το κείμενο, είναι ιδιαίτερα σημαντικός δεδομένης της ε, μεγάλης αναλογίας και αυξανόμενης των ανθρώπων που έχουμε μεταξύ των νέων που προέρχονται από τη μετανάστευση, κυρίως σε μερικές χώρες μέλη. Κλείνουν εδώ τα εισαγωγικά. Ανέφερα αυτά που λέτε, έτσι, τίποτα άλλο. Οπότε, ναι, θέλουμε κατευθυντήριες γραμμές, αλλά θέλουμε κατευθυντήριες γραμμές που να μπορούν να υλοποιηθούν με νούμερα ρεαλιστικές και να ξαναδούμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και που προς το παρόν κύριε Καλβεσαμπό με κάθε σεβασμό που σας οφείλω απέδειξαν την αποτυχία των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της απασχόλησης χρόνο το χρόνο δεκαετία μετά τη δεκαετία Κυρία Συγήτρια δεν σας ε, ζηλεύω αλλά καταλαβαίνω γιατί είσαστε απογοτευμένοι. Ευχαριστώ. Η κυρία Τσανόκα. Τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ναι, μετά από αυτήν την τόσο εντυπωσιακή παρέμβαση του κύριου Μαρτά, τι να πω. Εξακολουθώ εγώ να πιστεύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κοινωνική Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχομαι από μία από τις νέες χώρες μέλη, της Ανατολικής Ευρώπης που το 2004 ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά το 2007 είχαμε και άλλες δύο και άλλη μία αργότερα που εντάχθηκε. Ναι, είμαστε η Ευρώπη των 28 σήμερα. Και δεν με ικανοποιεί καθόλου η διαδικασία που ακολουθούμε και που οδηγεί σε μεγαλύτερη διαφοροποίηση ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς, τις πλούσιες χώρες και τις φτωχές χώρες, με μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν κτλ. κτλ. Ελπίζω πραγματικά ότι μπορούμε να πετύχουμε μία εναρμόνιση σε ένα κείμενο που να εγκρίνουμε οι περισσότερες πολιτικές ομάδες. Είπα και στην εισαγωγή μου ότι πρέπει να παρουσιάσουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τουλάχιστον υπάρχει μια ισχυρή πλειοψηφία. Έχουμε λοιπόν στη διαθεσή μας μια στέρεα βάση γι' αυτό, τον κοινωνικό πυλώνα, και ελπίζω ειλικρινά ότι θα καταλήξουμε σε ένα έγγραφο που θα είναι το κατάλληλο. Το πρόβλημα για μένα τώρα είναι πώς το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εδώ υπάρχουν πολλές αφιβολίες... για το κατά πόσο θα το κάνει. Παρ' όλα αυτά, εμείς πρέπει να κάνουμε τη δικιά μας τη δουλειά. Είμαστε εκλεγμένοι από τους λαούς μας Είμαστε εδώ αντιπροσωπεύοντας τα δικά τους τα συμφέροντα. Ο κόσμος θέλει περισσότερα κοινωνικά δικαιώματα. Και εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε εδώ εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σωστά. Θέλετε να προσθέσετε κάτι από αυτού. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που δίνετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο για να εξηγήσουμε. Πρώτα απ' όλα, οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση αυτή τη φορά εγκρίθηκαν ή τροποποιήθηκαν τέλος πάντων βάσει των ε, αρχικών αρχών. Ε, κάναμε δηλαδή πολύ προσεκτικά σύγκριση με τις αρχές και προσπαθήσαμε να δούμε πώς καλύτερα θα, σωματι... θα τις ενσωματώσουμε αυτές τις νέες κατευθυντήρες γραμμές. Είναι κάτι πολύ θετικό γιατί όπως ε, ξέρετε ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων ήταν κάτι που ήθελαν όλες οι χώρες μέλη. Άρα όλες οι χώρες το στηρίζουν. Τώρα, κι εμείς προσβλέπουμε σε συνεργασία με την εισηγήτρια και τους σκιώδες εισηγητές. Οπότε, εάν χρειάζεστε περισσότερες επεξηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαρίστως να ξανάρθουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Άλλος κανείς θέλει το λόγο. Όχι από ό,τι βλέπω. Καλώς. Οπότε, τώρα έχουμε κερδίσει χρόνο, ε. Τώρα θα έπρεπε Έχουμε 40 λεφτά μέχρι να μπορέσουμε να αρχίσουμε με την επόμενη έκθεση που πρόκειται για την ισορροπία ιδιωτική και επαγγελματική ζωής. Δεν ξέρω τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει εκπρόσωπος της Επιτροπής εδώ για την ισορροπία αυτή ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής μήπως. Για να αρχίζαμε τώρα. Θα διακόψουμε για λίγο και μετά θα περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και ιδιωτική ζωή για γονεί και ανθρώπου που φροντίζουν παιδιά. Yes, we hear now that there will be... Τώρα μόλις μας ενημέρωσαν ότι θα έρθουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε 7 λεπτά θα είναι εδώ. Οπότε 7 λεπτά διάλειμμα παρακαλώ.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

Κυρίε uh, uh, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ε, είμαστε βέβαια τώρα πάλι πληρείς, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τις καθυστερήσεις για ένα 20 λεπτό ακόμη. Θα προχωρήσουμε λοιπόν με το θέμα της ημερησίας διατάξεως, αλλά είμαστε και 20 λεπτά πριν από την προβλεπόμενη ώρα. Θα δώσω πρώτα τον λόγο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουν μάλιστα και οπτική παρουσίαση, όπως θα είδατε. Θα μας μιλήσουν για την εξισορρόπηση επαγγελματικού και προσωπικού βίου. Πρόκειται για τις Γενικές Διευθύνσεις Απασχόλησης και Δικαιοσύνης. Δύο χωριστές διευθύνσεις δηλαδή. Γενικές διευθύνσεις ακόμα καλύτερα. Εσείς πρώτα κύριε από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Πράγματι θα δούμε τα βασικά στοιχεία της δέσμης μέτρων της εξισορρόπησης επαγγελματικού ιδιωτικού βίου σε αυτή την παρουσίαση. Όπως ξέρετε είναι μέρος του κοινωνικού πυλώνα αυτή η διάσταση. Είναι μια απόκληση σε κάποιες από τις αναπομείνασες προκλήσεις που δεν έχουν ακόμη επιληθεί και βασική τομής πρωτοβουλίας είναι αυτά που καλύπτει η πρόταση οδηγίας και η ανακοίνωση της Επιτροπής. Όπως ξέρετε, τον Απρίλιο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων που υποστηρίχθηκε, εγκρίθηκε μάλλον στο τέλος του έτους. Ε, είναι ταχύε οι εξελίξει της κοινωνία μα στον επίπεδο τη εργασία, των δημογραφικών αλλαγών, τη ψηφιακή εξέλιξη και τη παγκοσμιοποίηση. Και αυτή ήταν η απόκρισή μα. Έχουν δημιουργηθεί νέες ευκαιρίες και δυσκολίες και ο πυλώνας έχει να κάνει με την εξασφάλιση δικαιωμάτων για τους πολίτες σε, αυτή, σε αυτές τις νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Θέλει να, να, να βρει μια νέα διαδικασία αναθέρμανσης του οικονομικού και κοινωνικού της οικονομικής και κοινωνικής πρόοδου και εδώ έχουμε τα βασικά στοιχεία των αρχών που θα διέπουν την εξορρόπηση ιδιωτικού και επαγγελματικού βία, βίου. Ε, όλα αυτά σχετίζονται με την πρωτοβουλία για την εκπαίδευση, για την ισότητα των φίλων, τις ίσες ευκαιρίες και την στήριξη της απασχόλησης. Αυτό έχει να κάνει με τα δικαιώματα, των, την υποστήριξη των γονιών και όσων έχουν υποχρεώσεις φροντίδας, την πρόσβαση σε ανάλογες υπηρεσίες καθώς και σε γονικές άδειες. Επίσης, οι διαθετήσεις θεώρησης για ε, άνδρες και γυναίκες είναι κάτι το σημαντικό. Οι ε, υποχρεώσεις φροντίδας επίσης παιδιών και ηλικιωμένων είναι κάτι που θα μας απασχολήσει. Τώρα να πω λίγα λόγια για τις βασικές προκλήσεις της πρωτοβουλίας για την εξισορρόπηση επαγγελματικού ιδιωτικού βίου κυρίως έχουν αλλάξει κυρίως οι συσχετισμοί εντό της ε, αγοράς εργασίας. Οι γυναίκες έχουν πλέον πολύ ψηλά προσόντα και τα εργασιακά τους δικαιώματα αυξάνονται. Όμως πέραν αυτών των θετικών αλλαγών οι, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας. Ξέρουμε ότι ο συνολικός δείκτης απασχόλησής τους είναι 12% κάτω από αυτών των ανδρών και είναι 18% σε μονάδες ε, μέτρησης της πλήρους απασχόλησης σε κάποιες χώρες. Μπορεί να φτάνει και υψηλότερα ποσοστά. Ιδίως αν μετρήσουμε και τις γυναίκες που απασχολούνται σε θέσεις ε, μερικής απασχόλησης. Επίσης για το χάσμα στις αμοιβέ φτάνει το 16% αν πάρουμε το μεσόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σχετικό με αυτό, ο ρόλος του γονέα και άλλες υποχρεώσεις φροντίδας δεν είναι σωστή η εξισορρόπηση που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γυναίκες περνούν διπλάσιο χρόνο στις υποχρεώσεις αυτές από ότι οι άντρες. Και περίπου σε όλα τα κράτη-μέλη με το μισθολογικό χάσμα έχουμε 9% γυναίκες με ένα παιδί που μπορεί να φτάσει και το 30% να απασχολούνται στο σπίτι. Ίσως δεν είναι τόσο γνωστό ότι ο ρόλος του γονέα για τους άντρες έχει την αντίθετη συνέπεια. Οι γονείς με ένα παιδί κάτω των 6 έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν δουλειά. Δηλαδή, ε, το ποσοστό απασχόληση ε, των ανδρών με ένα παιδί κάτω των 6 είναι 12% ε, σε κάποιε χώρε. Ω προς το σχεδιασμό πολιτικής υπάρχουν τρεις βασικές προκλήσεις που καλείται να καλύψει η δέσμοι και έχουν να κάνουν με την άνηση κατανομή των υποχρεώσεων φροντίδας. Πρώτα απ' όλα η ακατάλληλες γονικές άδειες και οι αδιάλακτες εργασιακές διευθετήσεις. Η έλλειψη δικαιωμάτων άδεια μπορεί να επηρεάσουν την απόφαση μια γυναίκα να μένει στο σπίτι ή να επιστρέψει στην αγορά εργασία αφού αναλάβει υποχρεώσει φροντίδα. Όμω η πρωτοβουλία θέλει να κοιτάξει κατά την διάθεση και προσφορά ε, πατρικής ε, γονικής άδειας για πατεράδες. Αυτό θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στην κατανομή εργασίας και φροντίδας μεταξύ ε, πατέρων καθώς και τις προοπτικές απασχόλησης αργότερα. Ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη που έχουν ε, συγκεκριμένο ε, μερίδιο άδεια για πατέρες και το έχουν στοχεύσει, ε, έχουν θετικά αποτελέσματα γιατί αναλαμβάνουν υποχρεώσεις οι άντρες και συνολικά έχουν υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης. Η έλλειψη άδεια και για την φροντίδα άλλων εξαρτώμενων μελών τη οικογένεια. Επηρεάζει και άντρε και γυναίκε σήμερα όπου δεν υπάρχουν ε, ε, ρήτρε για την ε, διθέτηση της φροντίδας γενικώ. Συνήθως το λογαριασμό των πληρώνουν οι γυναίκες και όχι οι άντρες. Και επειδή δεν υπάρχουν και διαλλακτικές εργασιακές διευθετήσεις, πάλι οι γυναίκες μένουν εκτός αγοράς εργασίας όταν αναλαμβάνουν υποχρεώσεις φροντίδας ή ζητούν ευέλικτε εργασιακέ συνθήκε. Χρειάζονται προσαρμοσμένα ωράρια, προσαρμοσμένες διευθετήσεις και ε, περισσότερο περιθώριο για να ε, εκτελέσουν τις υποχρεώσεις φροντίδας. Η δεύτερη συνέπεια από την άνηση κατανομή υποχρεώσεων φροντίδας μεταξύ άνδρων και γυναικών είναι η προσφορά φτηνών υπηρεσιών φροντίδας ε, είτε είναι για τα παιδιά είτε άλλες μορφής και η δυσκολία πρόσβασης για να υπάρξει ε, εφόσον δεν υπάρχει μόνο πρόσβαση σε τέτοιου είδου ε, υπηρεσίε, οι γυναίκε αναγκάζονται να μειώσουν το χρόνο που εργάζονται. Γνωρίζετε καλά του στόχου, καθώ και τι προβλέπει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων. Στόχο είναι να αυξηθεί περαιτέρω η πρόσβαση στην επίσημη φροντίδα παιδιών. Η έλλειψη επίσημων διευθετήσεων για το φροντίδα των παιδιών μπορεί να οδηγήσει πολλούς ενδεχομένως συγγενείς, κυρίως γυναίκες, να αναλάβουν το ρόλο του φροντιστή. Το πρόβλημα με τους εξαρτώμενους συγγενείς είναι μεγαλύτερο στην ηλικιακή ομάδα 50 έως 60 ε, ετών και μία στις έξι γυναίκες, μάλλον οι γυναίκες είναι έξι φορές πιο πιθανό να αναλάβουν ρόλο φροντιστή από ότι αναλόγως οι άντρες. η ελληπής ε, ισότητα κατανομής των υποχρεώσεων φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών επηρεάζει και τις, ε, οικονομικά, τις οικονομικές προσόδους μιας οικογένειας. Ε, κάποια κράτη βέβαια έχουν ε, φορολογικά κίνητρα με την ε, φορολογία, με τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τα νοικοκυριά όπου κάποιοι έχουν μία πηγή εισοδήματος σαν οικογένεια Εκεί δημιουργούνται κάποια φορολογικά περιθώρια που αποθαρρύνουν τους άντρες ή γυναίκες να μπουν στην αγορά εργασίας ή να αυξήσουν το ωράριο εργασίας τους. Υπάρχουν επίσης κάποια φορολογικά αντικίνητρα σε κάποια κάτι μέλη, ενώ μεγαλύτερος αριθμός κατών μελών έχουν κάποιο είδους αντικίνητρο που προκύπτει με το φόρο, ακόμη και αν υπάρχει επίδομα για τη φροντίδα των παιδιών. Συνολικά αυτά μεταφράζονται σε δυο λογιών κόστη, τα ιδιωτικά και τα δημόσια, διότι οι πολίτες, οι γυναίκες κυρίως έχουν λιγότερες ευκαιρίες διαδρομία. περισσότερη απειλή στην αγορά ε, απασχόλησης, ενώ οι άντρες αντιμετωπίζουν ε, δυσκολίε να συμφιλειώσουν ιδιωτικό και επαγγελματικό βίο, η μεγαλύτερη απειλή φτώχεια για τα παιδιά. Οι εταιρείε έχουν έλλειψη σε δεξιότητε, δυσκολία να κρατήσουν του εργαζόμενου, χαμηλότερη παραγωγικότητα και χαμηλότερη προσώπηση των γυναικών σε θέσει management, σε υψηλότερα κλιμάκια. Τα κράτη-μέλη και οι προπολογισμοί του πιέζονται λόγω της δημοσιονομικής ε, μη βιωσιμότητας και η οικονομία συνολικά πληρώνει το αντίτιμο της ανισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν εκτιμήσεις που λένε ότι φτάνουμε τα 370 δις ετησίως. 3% του ΑΕΠ. Είναι σημαντικό ποσό. Και μερικές ενιστώσεις όπως η κατασπατάληση δημοσίων πόρων, οι επενδύσεις και ούτω καθεξής δεν συμπεριλαμβάνονται. Η πρωτοβουλία για την εξισορρόπηση επαγγελματικού ιδιωτικού βίου έχει σκοπό να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες στο πλαίσιο της ανάκλησης της οδηγίας 2010 του του 2010 για να ξαναδούμε την ε, άδεια μετρότητας. Θα πρέπει να την ε, αναθεωρήσουμε με βάση τις νέες κοινωνικές εξελίξεις. Αυτή η πρωτοβουλία έχει σκοπό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχουν οι γυναίκε με την εκπροσώπησή του στην αγορά εργασία και με διαφορετικά ευρωπαϊκά εργαλεία που μπορεί να δώσουν ε, τη δυνατότητα στου γονεί και άλλου όσου ε, που μπορεί να έχουν υποχρεώσει φροντίδα να εξορροπήσουν τον επαγγελματικό και ιδιωτικό του βίο και να ενθαρρύνουμε την καλύτερη κατανομή υποχρεώσεων φροντίδα μεταξύ των ανδρών και των γυναικών. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει ένα συνδυασμό εργαλείων, πρόταση οδηγίας και μια ανακοίνωση της Επιτροπής. Τα βασικά στοιχεία της πρότασης οδηγίας που βασίζεται σε μια ευρύτερη προσέγγιση και τα εργασιακά δικαιώματα είναι η πρόβλεψη άδειας πατρότητας βάσει της οποίας θα μπορούν ε, οι πατέρες να παίρνουν 10 ημέρες άδεια ε, αμοιβόμενοι όπως και η άδεια στενίας η αναρωτική θα είναι μάλιστα υποχρεωτική τη στιγμή της γέννησης ε, ενό παιδιού αυτή η δεκαήμερη άδεια Επίση, η θέσπιση αυτού του δικαιώματο θα πρέπει να έχει θετικό αντίκτυπο στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία επίσης και μόχλευση. Θα προσφέρει μόχλευση για την ε, λήψη άδεια από τους άντρε. Στην Πορτογαλία, λόγω χάρη, όπου η άδεια πατρότητας έχει ενισχυθεί πολύ, εκεί 80% των πατέρων παίρνουν την άδεια πατρότητας και χρησιμοποιούν και τη γονική άδεια. Ενίσχυση τώρα Τη γονική άδεια είναι επίσης ε, σημαντικό στοιχείο τη πρότασης οδηγία. Η θεμελίωση δικαιώματος υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τέσσερις μήνες που μπορεί να πάρει αυτή την άδεια μέχρι τα 8 έτη του παιδιού του μπορεί να μεταφέρει τρεις μήνες στον άλλο γονέα και συνήθως μέχρι τώρα αυτό που ισχύει είναι ότι οι μητέρες παίρνουν το μερίδιο των πατέρων. Η πρόταση διατηρεί το τετράμινο που υπάρχει, αλλά το ενισχύει με μία αντιστάθμιση, τουλάχιστον στο επίπεδο της αναρωτικής άδεια και το δικαίωμα γίνεται μη ε, μεταβιβάσιμο από τον ένα γονέα στον άλλο. Οι γονεί κατόπιν αιτήματο μπορούν να πάρουν την άδεια με τρόπο διαλεκτικό ευελικτό μέχρι το παιδί να φτάσει τα 12 έτη του. Βλέπουμε λοιπόν όντω ότι στα κράτη-μέλη που έχουν στοχεύσει το, ένα σοβαρό μερίδιο τη άδεια για του πατέρε και τη γονική άδεια την προσφέρουν σε καλά επίπεδα, έχουν και περισσότερη λήψη αδειών από πατέρε καθώς και καλύτερα αποτελέσματα για τις μητέρες σε επίπεδο αποσχόλησης. Στη Σουηδία και τη Γερμανία, λόγου χάρη. Η πρόταση οδηγίας επίσης περιλαμβάνει διατάξεις για την άδεια των φροντιστών, για ε, όσους ασχολούνται με τη φροντίδα ατόμων της οικογένειας με σοβαρές παθήσεις, νόσους, ασθένειες ή με αναπηρίες εδώ δεν υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας. Ο εργαζόμενος μπορεί να πάρει άδεια για σύντομο χρονικό διάστημα για λόγους ανωτέρας βίας ή για επίγουσες οικογενειακές ανάγκες. Όπως βλέπετε δεξιά, προβλέπεται οι εργαζόμενοι φροντιστές να παίρνουν πέντε μέρες θυσίως, να παίρνουν αμοιβή τουλάχιστον στο επίπεδο της αναρωτικής και όταν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση Επίσης χρειάζονται και οι ε, ελαστικές διαθετήσεις ε, στην ε, εργασία. Το δικαίωμα αυτό θα θεμελιωθεί, θεμελιώνεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Τώρα οι γονείς μπορούν να ζητήσουν μειωμένες ή προσαρμοσμένες ώρες εργασίας βάσει και της γονικής άδειας. Η νέα πρόταση προβλέπει την δυνατότητα της μερικής εργασίας για όλους τους εργαζόμενους όλοι οι γονείς των παιδιών μέχρι τα 12, οι φροντιστές μπορούν να ζητήσουν Μπορούν να ζητήσουν προσαρμοσμένο ωράριο ή μειωμένο ωράριο ή ελαστική εργασία ή να τους προσφερθεί ελαστικότητα στο χώρο εργασίας. Ε, επιπλέον, η πρόταση προβλέπει προστασία για εργαζόμενους που θα ε, σκούν αυτά τα δικαιώματα. Αυτά είναι ίσως τα βασικά στοιχεία της πρότασης οδηγίας ή αδιαπατρότητας, κάτι που δεν προβλεπόταν ως τώρα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ή διατάξεις για τη γονική άδεια που πάνε πέρα από τις ισχύουσες διατάξεις όσα προβλέπονται για τους φροντιστές και την αδειά τους, κάτι που διευρύνει το πεδίο των τωρινών διατάξεων και οι ευέλικτε, οι ελαστικές διαθετήσει εργασίας που υπήρχαν ε, εν μέρη και στην ισχύουσα οδηγία προκειμένου να συμπληρώσουμε αυτήν την νομοθετική πρόταση, ε, η πρωτοβουλία περιέχει και μια σειρά από μη νομοθετικά μέτρα για να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη προκειμένου να πετύχουν καλύτερη εξισορρόπηση εργασιακού ιδιωτικού βίου. Αυτά τα παρουσιάζει η ανακοίνωση που είναι μέρος της πρωτοβουλίας. Υπάρχουν τρεις τομείς προτεραιότητες που ε, παρουσιάζονται εδώ συνοπτικά. Ο πρώτος έχει να κάνει με την, ε, τον οικογενειακό βίο και το συνδυασμό με, την, ε, με τις ελαστικές διευθυντήσεις ασφάλειας. Μετά η οδηγία με κάποια σημεία δράσης για να υλοποιηθεί καλύτερα η ισχύουσα νομοθεσία να βελτιωθεί η προστασία, η συλλογή δεδομένων και τα καινοτόμα προγράμματα. Και όπω ανέφερα προηγουμένω, η επίσημη βοήθεια, οι σχετικές υπηρεσίε και η αντιμετώπιση των οικονομικών αντικινήτρων είναι σημαντικέ δυσκολίες. Πρέπει να τα λύσουμε για να αντιμετωπίσουμε την ε, χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Άλλοι δύο τομεί λοιπόν πολιτική όπου θα πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση. Τα καλύπτει ανακοίνωση. Εκεί ε, αναπτύσσονται το ποιε είναι οι ελλείψεις των κρατομελών στους τομείς αυτούς και προτείνονται ε, βελτίωση της συλλογή ε, δεδομένων, λύτερη καθοδήγηση βάσει των συστάσεων προκύπτων και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και ανταλλαγή καλών πρακτικών, καθώς και επιπλέον χρηματοδότηση από το ΕΖΙΦ και το EFSI. Αυτά είναι τα κύρια συστατικά της πρωτοβουλίας εξισορρόπησης επαγγελματικού ιδιωτικού βίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Για να ολοκληρώσω, απλώς να πω ότι ενώ αναγνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετική κουλτούρα ως προς τα θέματα αυτά και διαφορετικά συστήματα, πιστεύουμε ωστόσο ότι η συνεργασία μας και η ανταλλαγή καλών πρακτικών θα μας επιτρέψει να επιζητήσουμε ε, επιτυχώς το στόχο εξισορρόπησης επαγγελματικού ιδιωτικού βίου. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Έχουμε εδώ ο εισηγητής Κιώδης. Περιμένουμε ακόμα. Η Γενική Διεύθυνση Just δεν είναι εδώ, από ό,τι φαίνεται. Thank you for being here. Please take... ευχαριστούμε. Καθίστε κι εσείς εδώ και έχετε το λόγο τώρα. Ή τέλος πάντων εσείς όπως θέλετε κατευθύνετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Έχουμε τα κύρια στοιχεία λοιπόν. της πρότασης αυτής, της πρωτοβουλίας αυτής. Να προσθέσω ότι αποτελεί μέρος του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων χρειαζόμαστε τη στήριξή σας. Έχουμε ήδη αρχίσει τη συζήτηση με τις χώρες μέλη και ο κύριος στόχος της πρωτοβουλίας αυτής στα πλαίσια του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων είναι να προχωρήσουμε περισσότερο στο τομέα της ισότητας, της ισορροπίας επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής γιατί σίγουρα έχει επιτευχθεί αρκετή πρόοδος μέχρι τώρα αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν περιθώρια για να γίνουν περισσότερα για δράση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρος, καλώς, ευχαριστούμε. Ο εισηγητής τότε έχει τώρα το λόγο για την απασχόληση, ο κύριος Κάσα του ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της. Και σας ευχαριστούμε που είσαστε και εδώ σήμερα. Η πρόταση αυτή λοιπόν είναι πολύ επίκαιρη αλλά είναι και αναγκαία προκειμένου να προχωρήσουμε στη διευθέτηση της ισορροπίας αυτής με μυδικέ άδειε, άδειε κλπ. προκειμένου να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ε, αλλαγές που διαπιστώνουμε στις κοινωνίες μας. Επίσης, θέλουμε να ε, μπορέσουν και οι άντρες να έχουν πιο ελαστικές συνθήκες εργασίας. Και αυτό το λέμε επειδή, όπω πολύ σωστά είπατε κι εσεί, δεν εκπροσωπούνται παρκώ στην απασχόληση οι γυναίκε. Θέλουμε λοιπόν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμφιλειωθεί η επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Το έργο μας πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτή τη νέα πραγματικότητα πολύ ισορροπημένα. Γι' αυτό και αξίζει να πούμε ότι πρόκειται για την πρώτη πρόταση που έχουμε από τον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που μόλις υπογράφηκε από τα τρία θεσμικά όργανα τον Νοέμβριο που μας πέρασε στη Σουηδία. Όπως είδαμε και από την παρουσίαση της πρότασης, εισάγει διάφορα νέα στοιχεία με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι ανομιλίε που έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν μέχρι τώρα για να πετύχουμε αυτή την ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική και επαγγελματική ζωή για τους γονείς και εκείνους που φροντίζουν οικείους τους. Υπάρχουν πολλά νέα στοιχεία λοιπόν τα οποία έχουν συζητηθεί με τους ενδιαφερόμενους. Είναι μια δουλειά που συνεχίζεται και πιστεύω ότι χρειάζεται παραπάνω διαβούλευση για να πετύχουμε αυτή την ισορροπία που θέλουμε. Κυρίως όμως χαίρομαι για το γεγονός ότι οι προτάσεις σας επικεντρώνονται και στην περίπτωση των ανθρώπων που φροντίζουν οικείους, οι οποίοι είναι όλο και περισσότεροι μεταξύ των συνανθρώπων μας. Όσον αφορά την άδεια πατρότητας, αυτό το οποίο προτείνεται πιστεύω ότι αποτελεί μία αυτή πρόοδο και είναι εφικτό ως λύση. Τώρα για να υπάρχει περισσότερη ευελιξία σε όλους τους εργαζόμενους γονείς πιστεύω ότι και αυτή είναι μια πολύ καλή πρόταση. Είμαι σίγουρος ότι με κάποιες μικρές αποχρώσεις θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την πρόταση αυτή που αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που υπάρχουν στην μέθοδο εργασίας και την ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή. Από την άλλη όμως περιμένω και κάποιους συμβιβασμού για αυτό που λέτε για τη μη μεταβίβαση των τεσσάρων μηνών ε, γονικής άδεια. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο με τους ενδιαφερόμενους για να βρούμε και εδώ τη σωστή ισορροπία που να μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά και για τις δύο πλευρές. Ένα άλλο στοιχείο που ίσως χρειάζεται παρατέρω συζήτηση είναι το θέμα της πληρωμής των αδειών αυτών σε επίπεδο αναρωτικής. Η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Από τις επαφές που είχα εγώ μέχρι τώρα με τους ενδιαφερόμενους φαίνεται ότι χρειάζεται περισσότερη διαβούλευση για να υπάρχει σωστή εκπροσώπηση όλων των απόψεων. Τέλος, υπογραμμίζω ότι θα προσπαθήσω και εγώ να δουλέψω για την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην εισαγωγή δικαιωμάτων για τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής από και από την άλλη μεριά την καλή λειτουργία των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων για παράδειγμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κάσα. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Μαρία Αρενά, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, με συγχωρείτε που καθυστέρησα κάπως, καμιά φορά είναι λίγο δύσκολο να συμφιλιώσουμε την επαγγελματική με την επαγγελματική μας ζωή, τρέχοντας από τη μία επιτροπή στην άλλη. Ευχαριστώ πάντως τον κύριο Κάσα για την παρουσίαση του ε, θέματος που είναι πράγματι τόσο σημαντικό, δηλαδή η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και προσωπικού βίου. Έχει γίνει μια μελέτη στην Γαλλία που δείχνει και αυτή νομίζω μπορεί να ισχύει και για το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, 57% των μισθωτών σήμερα αντιμετωπίζουν δυσκολίες ακόμα και για τα απλά γραφειοκρατικά θέματα. 50% δεν προλαβαίνουν τα οικιακά και από αυτά 16% δεν προλαβαίνουν καν να ασχοληθούν μετά του σπιτιού. Χρειάζεται λοιπόν απελευθερωθεί χρόνος, δύσκολο αυτό για την πλειοψηφία των προσώπων αυτών, 51% των μισθωτών λένε ότι δεν έχουν καν χρόνο για να περάσουν με τους οικείους τους και 40% δεν προλαβαίνουν να έχουν προσωπική ζωή εκτός εργασίας. Γι' αυτό ρωτώ, στην πραγματικότητα σκοτωνόμαστε στη δουλειά για να δουλεύουμε ή δουλεύουμε για να ζήσουμε καλύτερα. Εγώ προτιμώ την δεύτερη υπόθεση, δηλαδή να εργάζεται κανείς για να μπορέσει να βελτιώσει την ζωή του. Νομίζω αυτός πρέπει να είναι ο στόχος που θα πρέπει όλοι να επιδιώκουμε. Ε, μέσα στα πλαίσια αυτά, πρώτα επιθυμώ να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάληψη της πρωτοβουλίας. Έχουμε ζήσει ήδη από την αρχή της θητείας το δράμα αυτό, δηλαδή την εγκατάληψη της οδηγίας για την μητρική άδεια. Και λέω δράμα διότι ήταν μια θαυμάσια εργασία η οποία έχει γίνει και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δυστυχώς όμως λόγω έλλειψης βουλήσεως στο Συμβούλιο προφανώς ήταν δύσκολο να προχωρήσουν το Συμβούλιο δηλαδή στο θέμα αυτό. παρόλα αυτά όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέρχεται, αναλαμβάνει πρωτοβουλία και θεωρώ ότι η Αρμοδία Επίτροπος αντιλαμβάνεται ποια είναι η δυσχέρεια σήμερα. Όχι όμως μόνο μια δυσχέρεια για την συμφιλίωση των δύο αυτών πτυχών της ζωής, αλλά και συμφιλίωση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων και της ισορροπίας ανδρών και γυναικών στην εργασία. Επομένως, το, ο φάκελος αυτός έρχεται να πάρει χέρι με χέρι και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Πάνω από 50% των εργαζόμενων δεν αισθάνονται καλά στη δουλειά τους. Επομένως η παραγωγικότητά τους δεν θα είναι βεβαίως αυτή που θα ανέμενε κανείς. Εάν οι γυναίκες οι οποίες έχουν προσόντα, έχουν διπλώματα, δεν μπορούν να εισέλθουν στον χώρο της εργασίας, στην ουσία πετούμε τα λεφτά μας στα σκουπίδια. Δηλαδή πληρώνουμε για την εκπαίδευση των γυναικών αυτών, η οποία εν τέλει δεν αποδίδει. Ε, να σας δώσω ένα νούμερο. Μία γυναίκα με τρία παιδιά, η συμμετοχή δηλαδή των γυναικών που έχουν τρία παιδιά στην απασχόληση μειώνεται πάνω από το 50%. Ενώ ένας άνδρας τρίτεκνος η συμμετοχή του φτάνει στο 80%. Για φανταστείτε τα στερεότυπα μέσα στα οποία ζούμε σήμερα. Άρα χρειάζεται ανάληψη δράσης. Υπάρχει η Ένωση των Οικογενειών μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΚΟΦΑΣ που ανέλαβε την πρωτοβουλία, μάλλον που δέχεται την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τρεις πυλώνες. Πρώτον, υποχρεωτική πατρική άδεια 10 πληρωμένων ημερών για να ξαναμπούν οι άνδρες, οι πατεράδες δηλαδή, μέσα στον οικογενειακό βίο, διότι έχουν και ρόλο να παίξουν. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι αν αυτή η άδεια δεν είναι υποχρεωτική, η κοινωνική πίεση από την επιχείρηση θα οδηγήσει να μην την πάρουν και αν δεν είναι πληρωμένη, χάνει πολλά ο πατέρας ε, από το εισόδημα της οικογένειας. Άρα η βούληση να υπάρχει υποχρεωτική άδεια που να πληρώνεται. Δεύτερο, ε, γονική άδεια. Θα χρειαστεί βεβαίως να ασχοληθούμε περισσότερο με την δυνατότητα μεταφοράς. Σήμερα πάντως η γονική άδεια λαμβάνεται από το 2,7% των ανδρών στην Ευρώπη. Όταν μιλούμε για γονική άδεια, 2 και λίγο παραπάνω της εκατό των ανδρών παίρνει τη γονική αυτή άδεια. Θα προσθέσουμε τώρα και τη δυνατότητα μεταφοράς, δηλαδή ακόμα περισσότερες γυναίκες θα την πάρουν τότε, διότι το στερεότυπα είναι ότι εφόσον γίνεται να μεταφερθεί, η άδεια αυτή μεταφέρεται στις γυναίκες, είναι προφανές. Γιατί λοιπόν να γίνει, γιατί λοιπόν να πάρει κανεί την άδεια αυτή. Είναι σημαντικό να επανέλθουν οι άνδρες στη γονική άδεια. 2% μου φαίνεται ότι είναι, είμαστε πολύ μακριά από την ε, εξίσωση σε θέματα γονικής άδεια. Και επίση η αμοιβή τη γονικής άδεια. Γιατί είναι σημαντική η αμοιβή, διότι αν δεν γίνει αντιλαμβάνομαι το επιχείρημα ορισμένων που λένε ότι όντω επιβαρύνει οικονομικά τι επιχειρήσει. Είναι και ένα λόγο που θεωρώ ότι περιλαμβάνεται, για τον οποίο θεωρώ ότι περιλαμβάνεται μια πρόταση στην πρωτοβουλία τη Κομισιόν να μπει ένα σύστημα αλληλεγγύη. Ε, μέσα από ένα σύστημα δηλαδή κοινωνική προστασία και κοινωνική αλληλεγγύη που να πληρώνει αυτή την αμοιβή και να μην αναλαμβάνει ατομικά η κάθε επιχείρηση. Καταλαβαίνω βέβαια το επιχείρημα του Κάσα που λέει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναλαμβάνουν μεγάλο βάρος εάν γίνεται καθαρά ατομικά η πληρωμή τη άδεια. Χρειάζεται λοιπόν ένα στοιχείο αλληλεγγύης. Επανέρχομαι όμω στην αμοιβόμενη άδεια. Εάν δεν αμοιβόμενη τι θα γίνει. Σήμερα δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Τα ίδια τα νοικοκυριά πληρώνουν τελικά τη μείωση του χρόνου εργασίας και ιδίω οι γυναίκε, Διότι επειδή δεν αμείβεται η άδεια και επειδή υποχρεωμένε να κάνουν τα πράγματα αυτά, φτωχαίνουν τελικά, διότι είναι υποχρεωμένε να εγκαταλείψουν την αμοιβόμενη εργασία. Όταν λοιπόν μιλούμε για αμοιβόμενη εργασία, κατανοώ τα επιχειρήματα των επιχειρήσεων, αλλά από την άλλη μεριά ακούω και τα επιχειρήματα των γυναικών, οι οποίε ζουν και κάτω από το κατόφλι τη φτώχεια. Και μάλιστα όταν είναι μονογονικέ οι οικογένειε και είναι υποχρεωμένε να κρατούν τα παιδιά του και δεν υπάρχει άλλο να τα αναλάβει. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει απολύτω καμιά αλληλεγγύη και εκεί το άτομο πληρώνει τελικώ. Βεβαίω υπάρχει το επιχείρημα, ναι, ποιο πληρώνει. Εγώ λέω χρειάζεται επιλογή προτιμώ να υπάρχει ένα πρώτο επίπεδο αλληλεγγύης που θα είναι η επιχείρηση αντί να μην υπάρχει, να μην υπάρχει απολύτως κανένα επίπεδο αλληλεγγύης που είναι τελικώς η μάνα αυτή, η μαμά είναι αυτή η οποία αναλαμβάνει το βάρος των παιδιών και η οποία καταλήγει να φτωχύνει επειδή υπάρχουν τα παιδιά. Και μετά μιλούμε για ε, γεννήσεις πάρα πολύ χαμηλές για γεννητικότητα πάρα πάρα πολύ χαμηλή. Βεβαίως χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ευημερία της οικογένειες ώστε να ανέλθει και, το, και η γενετικότητα. Τέλος, τα πρόσωπα που προσφέρουν βοήθεια όσοι φροντίζουν. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε τον κοινωνικό αυτό ιστό στην Ευρώπη που βασίζεται όσο ολόκληρη ήπειρο το στοιχείο αυτό, θα πρέπει να μπορεί να διατεθεί χρόνος σε άλλο πρόσωπο της οικογένειας που διέρχεται μια κατάσταση καμιά φορά δραματική. Ασθένεια, άλλες δυσκολίες πρέπει να είναι δυνατόν να του προσφέρουν τα, οι άλλοι εκεί κάποιο χρόνο. Και εκεί πρέπει λοιπόν να είναι αμοιβόμενη αυτή η δραστηριότητα και γι' αυτό ευχαριστώ την πρωτοβουλία, για την πρωτοβουλία την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίω και είμαστε στη διάθεση του εισηγητού για να συζητήσουμε κάποια διαχείριση διότι η πρωτοβουλία αυτή είναι μια πρωτοβουλία η οποία τιμά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Βεβαίω και την Κομισιόν Juncker και το Συμβούλιο Υπουργών, αλλά βεβαίω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δείξει η Ευρώπη το κοινωνικό της πρόσωπο για το οποίο μιλήσαμε στο Γκέτενμπουργκ αλλά και αλλού. Κοινωνικό πρόσωπο απέναντι στους απασχολούμενους, στις επιχειρήσεις, στις μητέρες και στους υπολείπους. Θα συνεργαστούμε πολύ επικοδομητικά με τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, Ευχαριστούμε. Παρακαλώ κύριε Στάνσκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ βεβαίω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίω είναι σημαντικό να δοθεί περισσότερος χώρος στις γυναίκες και στην απασχόληση αλλά και στις οικογένειες διότι όταν μιλούμε για την πατρική άδεια και τα σχετικά Εν τέλει αυτό που ενδιαφέρει είναι οι, τα μέλη της οικογένειας να μπορούν να περνούν περισσότερο χρόνο μεταξύ τους. Δεν μιλούμε μόνο για αμοιβόμενους, για μισθωτούς πατεράδες και δεν είναι μόνο το θέμα αυτό, είναι να μπορούν να έχουν κοινό χρόνο. Εδώ νομίζω πρέπει να γίνει μια παρατήρηση ότι δηλαδή εδώ οφείλουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε τρόπο ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν και τα συμφέροντα των οικογενειών αλλά και αυτά των ε, εργοδοτών. Εγώ ε, δουλεύω πολύ με αναπήρους ανθρώπους και νομίζω ότι η φροντίδα των αναπήρων και οι άνθρωποι που προσφέρουν τη φροντίδα αυτή είναι πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερη σημασία. Έχουμε πολλούς ατομικούς ε, φροντιστές εντό εισαγωγικών που υποχρώνονται να καταλήξουν εν μέρη την επαγγελματική τους απασχόληση και εντελώς. Και γι' αυτό είναι αναγκαίο να βελτιώσουμε την θέση τους. Άλλωστε, και για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι που έχουν μια ανεξάρτητη επαγγελματική ε, απασχόληση πάλι αυτοί δεν μπορούν να δεν έχουν την αναγκαία ευκαμψία. Θα συνεργαστώ και εγώ βεβαίως με τον εισηγητή. Thank you. Ευχαριστούμε. Η Ραντεβέμπε δεν είναι εδώ, από ό,τι βλέπω. Η Τάνια Κονζάλες Πένιας, παρακαλώ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε προκειμένου να έχουμε ανταλλαγή απόψεων μαζί τους για την πρόταση αυτή οδηγίας. Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση η οποία δημιουργεί πολλές προσδοκίες στην ευρωπαϊκή κοινωνία και στις οικογένειες. Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία πάνω στο οποία πρέπει να δουλέψουμε. Όμως, κατά τη γνώμη μας, ξεκινάμε από ένα λάθος σημείο κίνησης. Δηλαδή για χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προχωράει σε μεταρρύθμιση της οδηγίας για τη μητρότητα και για μας το σωστό θα ήταν όλες τις υπάρχουσες οδηγίες να τις βάλουμε μαζί σε μια νέα. Γιατί το θέμα είναι η ανακατανομή ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες των όσων φροντίζουν παιδιά, οικείους κτλ. Πάνω από 50% είπαμε είναι οι γυναίκες αυτές που αναλαμβάνουν αυτά τα καθήκοντα και οι άντρες παίρνουν τις άδειε που τους αντιστοιχούν μόνο εφόσον αμείβονται πάνω από το 80% για αυτές. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο το πώς θα γίνει η ανακατανομή για να υπάρχει ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η κατανομή που δεν είναι καθόλου ισότιμη σήμερα αν δεν επιτευχθεί, σίγουρα οι γυναίκες πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να ενταχθούν και πάλι στην αγορά εργασίας. Όταν μένουν τόσα χρόνια εκτός αγοράς εργασίας, είναι πολύ πιο δύσκολες για αυτές να επαναδεχτούν. Αναφέρονται μόνο η γονική άδεια, η συμφιλίωση οικογενειακή επαγγελματική ζωή, δεν είναι πράγματα που φτάνουν. Συγκεκριμένα, τι μας απασχολεί. Ναι, στο να μην μεταβιβάζεται η άδεια, αλλά για την άδεια μητρότητας οι 10 ε, μέρες δεν προβλέπουν υποχρέωση. Δύο εβδομάδες δικαιούνται οι γυναίκες Όσον αφορά τη γονική άδεια για τα 12 πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού, είναι δύσκολο. Τι γίνεται με αυτή τη δυνατότητα. Συνήθως οι γονείς την παίρνουν αυτή την άδεια όταν είναι μωρά τα παιδιά τους και χρειάζονται κάποιον 24 ώρες το 24 ώρο δίπλα τους. Οπότε φοβάμαι ότι πάλι και αυτό θα πέσει στους ώμους των γυναικών. Εκείνες δηλαδή πάλι θα ασχολούνται με τα μωρά τους πρώτους χρόνους της ζωής τους. Από τα στοιχεία που έχουμε, οι άντρες παίρνουν την άδεια όταν αμείβονται, όπως είπαμε, 80% τουλάχιστον. Οπότε η αμοιβή είναι ζωτική σημασίας και θα πρέπει να δίνεται κατά 100% και όχι μόνο 80%. Κάτι άλλο που μας απασχολεί είναι το θέμα της ευέλικτης εργασίας. Είναι θετική αυτή η ιδέα της ελαστικής εργασίας. Δεν αναφέρεται τίποτα όμως για τις μονογονικές οικογένειες. Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να γίνεται τέτοια μνήμα. Και αυτές οι περιπτώσεις μονογονικών οικογενειών να μπορούν να επιλέξουν ένα τρίτο πρόσωπο να επωφελείται από τις άδειε αυτές που προβλέπονται για το δεύτερο γονέα. Και το θέμα της οικογένειας τώρα, ποια είναι αυτή η έννοια, πώς ορίζεται η έννοια αυτή, νομίζω πολύ αυστηρά ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία. Θα έπρεπε λοιπόν η έννοια οικογένεια να είναι ευρύτερη και στην περίπτωση των φροντιστών θα έπρεπε ο άνθρωπος ο οποίος έχει ανάγκη τη φροντίδα να επιλέξει αυτός ποιος θα το φροντίζει. Γιατί μπορεί να μην θέλει να είναι ο συγγενής του, να προτιμάει να είναι ένας φίλος του. Ε, κάποιος άλλος, οπότε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα επιλογής από αυτόν που έχει ανάγκη τη φροντίδα. Κατά τα άλλα, εντάξει, είναι θετική η πρόταση, εννοείται, και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να τη βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε κυρία Σντάνοκα. Πρόεδρε, Με ενθουσιασμό διαβάσαμε την πρόταση της Επιτροπής. Ήμουν συνεισηγήτρια του ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου που είχε τον τίτλο «Δημιουργώντας συνθήκες στην αγορά εργασία που να είναι ευνοϊκές για την εξισορρόπηση επαγγελματικού ιδιωτικού βίου». Εγκρίθηκε τον ε, Σεπτέμβριο του 2016 με δύο εισηγήτριες. Εμένα από ε, την Επιτροπή ε, Απασχόλησης και την κυρία Μπλινκεβιτσιούτα από την Επιτροπή Γυναικών. Ε, η σύνταξη αυτού του κειμένου ήταν ο καρπός πολλών συζητήσεων που φαίνεται ότι θα επαναλάβουμε και τώρα. Για την γονική άδεια, τα μεταβιβάσιμα ή μη δικαιώματα, μια άλλη πρόταση που επεψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο ήταν τα μερικώς μεταβιβάσιμα δικαιώματα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος να μην μπορεί να μεταφερθεί. Και άλλα αλληλένδετα προβλήματα. Εδώ απλώς να πω την θέση της ομάδας μου. είναι ότι θα συνεργαστούμε με τους κοιόδης εισηγητές της Επιτροπής Γυναικών και μετά από την ε, ε, διαβούλευση με μια σειρά από μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Είμαι βέβαια και, ότι και ο κύριος Κάζα είχε επίσης τέτοιου είδους ε, συζητήσεις. Θα πρέπει να πω ότι η άδεια μητρότητα. έμεινε ως είχε, αλλά ξέρουμε πόσα από πόσα προβλήματα πέρασε. Τώρα η πρόταση για την άδεια πατρότητας δεν μας αρέσει. Δεν είναι καλό αυτό με την αποζημίωση σε επίπεδο αναρωτική. Διαφέρουν πολύ αυτά από μια χώρα στην άλλη. Σε κάποιε υπάρχει το ελάχιστο 40% του μισθού και σε κάποιε όχι. Θέλαμε λοιπόν να το συζητήσουμε και να προτείνουμε κάτι παραπάνω. Υψηλότερο επίπεδο. 60 ή 80% τη κανονική αμοιβή. ως προς την άδεια, την γονική άδεια, το βασικό θέμα συζήτηση θα είναι το μεταβιβάσιμο. Κάποιοι θέλουν να μην υπάρχει καμία δυνατότητα μεταφοράς της γονικής άδειας από ένα στον άλλο. Πρέπει όμως να βρεθεί ένα συμβιβασμός. θα επεξεργαστούμε τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά. Σε ό,τι αφορά την αποζημίωση, οι παρατηρήσεις μου για την αδιαπατρότητα ισχύουν και εδώ. Το επίπεδο της αναρωτικής δεν είναι αρκετό, ιδίω για ορισμένα κρατημέλη. Εδώ θα θέλαμε να εισάγουμε και τους μόνους γονείς και ειδικέ προϋποθέσεις για αυτούς. Είναι ε, αμέλημα, είναι ε, παράβλεψη της, ε, αυλεψία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν ε, καλύπτει το θέμα αυτό ξεχωριστά. Οκτώ μήνες λοιπόν άδεια με δυνατότητα του μόνου γονέα να μοιραστεί την άδεια με άτομο της επιλογής του. Είτε συγγενή, είτε καταχωρη... καταγεγραμμένο μέλος ή όχι της οικογένειας, κάποιο γείτονα. Ιδιαίτερη κατάσταση αυτών των, αυτή των μόνων γονέων Πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν και αυτούς με τις μονογονεϊκές οικογένειες. Και να μην παρατάμε τις γυναίκες μόνο στην τύχη τους όπως είπε η κυρία Ρενά. Η άδεια των φροντιστών. Είναι πολύ θετικό αυτό το νέο στοιχείο που περιλαμβάνεται ε, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη έχουμε ε, προεξαγγείλει ε, ότι το περιμένουν οι πολίτες και βεβαίως το πενθήμερο μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως πιλωτικό πρόγραμμα. Ελπίζουμε ότι θα αναπτυχθεί στο μέλλον. Ναι. Και για τις ελαστικές διευθετήσεις στην εργασία. Πολύ καλές προτάσεις αλλά να θεμελιώσουμε, να προβλέψουμε και δικαίωμα, να θεσπίσουμε δικαίωμα να επανέλθει ο εργαζόμενος στο 100% της εργασίας του, όταν το επιθυμεί. Αυτά λίγο πολύ από πλευράς μας εν ώψη των συζητήσεων και διαβουλεύσεων με τον εισηγητή. Ευχαριστούμε. Με συγχωρείτε που το πω. Προσπαθήστε όμως να είστε πιο συνοπτικές και συνοπτικοί. Δεν έχουμε άπειρο χρόνο ώστε δεν θα έχουμε χρόνο να ομιλήσετε όλες και όλοι εάν ε, μακρηγορείτε. Η Λάουρα δεν είναι εδώ, της ομάδας EFTD. Ζουέλ Μιλάν από το ENF, Ευρώπη των Εθνών. Ήρθαμε κάποια καθυστέρηση διότι ήμουν σε άλλη επιτροπή και δεν μπόρεσα να ακούσω την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, έχοντας δει την έκθεση, αντιλαμβάνομαι προς ποια κατεύθυνση κινούμεθα αυτή την απίστευτη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταλήξει σε ισότητα ανδρών και γυναικών ακόμα και σε κάτι τι που καταρχήν φαίνεται τέλος πάντων να δείχνει ότι η ε, εργασία ελευθέρωσε τη γυναίκα και εξυπηρέτησε τον άνδρα. Εγώ έρχομαι σε ένα σημείο πολύ ιδιαίτερο της δύσκολης ισορροπίας για μια γυναίκα που εργάζεται ή έναν άνδρα που εργάζεται ανάμεσα σε μια επαγγελματική ζωή, προσωπική ζωή και μια τρίτη που είναι αυτή να ασχοληθεί με τους γονείς ή με ένα παιδί το οποίο έχει ένα βαθμό εξάρτησης. Είναι πολύ οδυνηρές ε, οι καταστάσεις αυτές και εκεί βεβαίως οι άνθρωποι που φροντίζουν τα πρόσωπα αυτά θέλουν να διατηρήσουν και μια επαγγελματική και προσωπική ζωή. Πολύ δύσκολο αυτό και δεν μπορεί να διευκολυνθεί με κείμενα οδηγιών ή κανονισμών κλπ. Σε κάθε χώρα μέλος θα πρέπει να θεσπιστεί νομοθεσία που θα επιτρέπει να χορηγηθεί βοήθεια είτε με ανάληψη βεβαίω και χρηματοδοτική, τεχνική και ανθρώπινη ε, το, το έργο των φροντιστών και αυτών που έχουν βαριές οικογενειακές υποχρεώσεις σε συνθήκες που δεν είναι πάντοτε και ορατές για να μπορούν να διατηρήσουν μια επαγγελματική δραστηριότητα. Δεν είναι ζήτημα των εργοδοτών αυτό πέρα από ένα απλό σχετικά πλαίσιο που θα είναι μια γονική άδεια ή μια, ε, μια άδεια του γιού ή της θυγατέρας. Και θα πρέπει το πλαίσιο αυτό να είναι τέτοιο που να επιτρέπει σε κάθε χώρα μέλους να ε, προβλέπει τέτοιε ρυθμίσει και ιδίω λόγω τη γύρανση του πληθυσμού για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να παραμένουν στα σπίτια του, αυτοί που έχουν ανάγκη δηλαδή. Κάθε πρόταση ευκαμψία ενό απλού πλαισίου που να επιτρέπει την διασύνδεση των δύο δραστηριοτήτων, δηλαδή επαγγελματικών δραστηριοτήτων και οικογενειακών δραστηριοτήτων που ε, βαραίνουν βεβαίω, δεν είναι δυνατόν όμως οι ε, άδειε αυτές να υπερβαίνουν κάποια διάρκεια που θα εμποδίζουν τους εργοδότες να ε, ε, διευθύνουν σωστά τις επιχειρήσεις Ευχαριστώ. Τώρα, ακούμε τη Γενική Διεύθυνση, ακούστε τη Γενική Διεύθυνση ε, Απασχόλησης και Δικαιοσύνης. Τώρα ακούσαμε και τους σχετικούς ε, εισηγητέ και συντονιστές, τώρα ερχόμαστε σε αυτού τη επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της. Πρέπει να πω ότι είναι μια σπάνια ευκαιρία όπου ένα θέμα για την αγορά εργασίας ρυθμίζεται με επιχειρήματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα της γυναίκας. Οπότε πρέπει να εκτιμήσουμε αυτή την ευκαιρία. Και είναι αλήθεια ότι η συμφιλίωση των ρόλων είναι μια δυσκολία για τις γυναίκες. Μια γυναίκα με παιδιά έχει πολλά προβλήματα να συμφιλιώσει την οικογενειακή με την επαγγελματική της ζωής και είναι θέματα που θεωρούμε ότι δεν αφορούν τους άντρες. Οπότε είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόταση για τα δικαιώματα των γυναικών επιτέλους και οι γυναίκες ήθιστε να είναι εκείνες υπεύθυνε για τις οικογένειές τους αλλά χωρίς να έχουν ένα εισόδημα όταν ασχολούνται με τα παιδιά τους ή με τους οικείους τους. Οπότε είναι υποχρεωμένες να εργαστούν. Συνεπώς έχει κάποια ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να τους επιτρέπει να εργάζονται και να μην έχουν όλες αυτές τις δυσκολίες να αντιμετωπίσουν. Μέχρι τώρα δεν έχουμε μιλήσει πολύ για τις λεπτομέρειες. Πάντως συζητήσαμε το θέμα της μη μεταβίβασης των δικαιωμάτων της άδεια. Είναι ένα πρόβλημα αυτό και γιατί, γιατί οι άντρες και οι γυναίκες έχουν διαφορετικές θέσεις στην αγορά εργασίας. έχουν ε, διαφορετικά δικαιώματα, οπότε δεν είναι η ίδια κατάσταση. Κάποιος άντρας που έχει παιδιά θεωρείται από τον ε, εργοδότη του σαν κάτι θετικό, γιατί θεωρείται ότι είναι ένας άνθρωπος πιστός, οικογενειάρχης, σοβαρός. Ενώ μια γυναίκα που έχει παιδιά δεν ε, της πιστώνεται αυτό σαν κάτι θετικό, γιατί θεωρείται ότι θα μπορεί να απασχοληθεί λιγότερο με τη δουλειά της και περισσότερο με τα παιδιά της ίσως. Οπότε είναι θέμα νοοτροπίας, είναι θέμα πώς αντιλαμβανόμαστε τον κάθε ρόλο του άντρα ή της γυναίκας. Θα έπρεπε τα ίδια κριτήρια να ισχύουν και για τους άντρες και τις γυναίκες και να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε οι άντρες να χρησιμοποιούν τις ευκαιρίες αυτές, τις άδειε αυτές. Τότε θα αλλάξει και η αντιμετώπιση στην αγορά εργασίας και θα είναι πιο δίκαια απέναντι στις γυναίκες. Και κοινωνικά είναι πολύ σημαντικό και για τις οικογένειες γιατί ένας άντρα ο οποίος προσέχει τα παιδιά του και ασχολείται με αυτά είναι μια καινοτομία και οι οικογένειες και τα παιδιά χρειάζονται τους πατεράδες τους. Μην ξεχνάμε ότι αν προσφέρουμε μία άδεια πατρότητας, ε, τότε η αξία αυξάνει στην αγορά εργασίας, γιατί θεωρείται ότι υπάρχει μεγαλύτερη ισότητα. Τέλος, η συνεργασία μας πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά για την πρόταση αυτή. Υπάρχουν κάποια ζητήματα προς επίλυση ακόμα, όπως αυτό που σας είπα, της μη ε, μεταβίβασης. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Για από τη μια μεριά λέμε ότι είναι σημαντικό οι άντρε να έχουν ανεξάρτητα δικαιώματα για τις άδειέ τους. Από την άλλη λέμε ότι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε κοινέ ε, προδιαγραφές και να μπορούν ίσως κάποιοι γονείς να παίρνουν τα παιδιά μαζί τους ε, εκεί που δουλεύουν. Σε κάποιες χώρες ισχύει αυτό, υπάρχει αυτό το δικαίωμα. Και μπορούν μερικές φορές συγχρόνως οι γονείς να παίρνουν τη γονική τους άδεια. Αν δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, τότε δεν μπορεί να γίνει αυτό να μπορούν συγχρόνως να έχουν ε, γονική άδεια γονείς. Πάντως Παρόλο που είναι φιλόδοξη η πρόταση αυτή, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές και αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γιαγκέριος έχει το λόγο που αντικαθιστά η κυρία Βιτσκεβισιούτε. Όχι, δεν ε, πρόκειται να την αντικαταστήσω εδώ. Για τους σοσιαλιστές μίλησε ήδη Μαρία Ρένα και εξήγησε ποια είναι η θέση της ομάδας μας. Εγώ ζήτησα το λόγο για να διευκρινίσω τρία ζητήματα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω να μου δίνετε την ευκαιρία γι' αυτό. Φυσικά Μιλάτε εκ μέρους της Επιτροπής Γυναικών, έτσι. Όχι. Ωραία. Τότε πρέπει να περιμένετε. Εσείς τότε. Εγώ δεν ε, συμμετείχα, έτσι καλλιώς δεν σκόπευα να είμαι εκπρόσωπος της Επιτροπής Γυναικών εδώ. Απλώς υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να σκεφτούμε. Η συμφιλίωση της επαγγελματική και της προσωπικής ζωής έχει να κάνει με τα δικαιώματα, τις άδειε κλπ. Όμως εγώ θα σας δώσω ένα στοιχείο εδώ, το οποίο είναι σημαντικό και ευχαριστώ την Επιτροπή για την πρόταση κειμένου της. Θα σας μιλήσω για την οικονομική πτυχή. Το Γαλλικό Παρατηρητήριο για την Οικονομική Συγκυρία ολοκλήρωσε μια έρευνα στους Γάλλους εργοδότες για όλες τις κατηγορίες και τους ρώτησε, θα θέλατε να έχετε περισσότερες ευθύνες εκεί όπου δουλεύετε, στους εργαζόμενους, έτσι. 78% των Γάλλων εργαζομένων, είτε άντρες είτε γυναίκες, απάντησαν όχι. Και το επιχείρημα ήταν ο φόβος ότι αν αναλάβουν περισσότερες ευθύνες στην επιχείρησή τους θα ζημίωνε ακριβώς την ισορροπία αυτή που έχουν πετύχει ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή. Και πολλοί εργοδότες ανησυχούν γι' αυτό. Άρα πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι και οικονομικό ζήτημα να πετύχουμε αυτή την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή. Και σας διαβεβαιώ, δεν κάνω λάθος, οι επόμενες γενιές, οι νέοι είναι πολύ πιο μακριά από εμά από αυτό το ιερό της καριέρας, της ζωής τους και δίνουν περισσότερη σημασία σε μια πιο ισορροπημένη οικογενειακή ζωή. Και εγώ τους λέω και πολύ καλά κάνουν. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος και δεν είναι εδώ. Η κυρία Μπέτρης Πεσέρα Παρεχέ δεν είναι εδώ, ούτε και αυτή με Κώστα... Κυρία παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την Επιτροπή για την ενημέρωση. Έχουμε μπροστά μας ίσως ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Εκείνο της οδηγίας και της στρατηγικής για την ισορροπία προσωπική και επαγγελματικής ζωής. Για το θέμα αυτό Δουλέψαμε πέρσι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της σύνταξης της έκθεσης πρωτοβουλίας που υιοθετήθηκε αλλά μάλλον δεν εισακούστηκε από την Επιτροπή αν κρίνω από το περιεχόμενο της οδηγίας. Με λύπη μου διαπίστωσα πως η πολύ διαφημιζόμενη νέα πρόταση οδηγίας η οποία θα ερχόταν να καλύψει εντός εισαγωγικών την την απόσυρση της νέας οδηγίας για την άδεια μητρότητας είναι δυστυχώς πολύ κατώτερη των προσδοκιών. Το χειρότερο όμως είναι πως αντί να ρυθμίζει τις αντιφατικές πολιτικές της Ένωσης και να καλύπτει τα κενά σε ό,τι αφορά τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών της, και τι με αυτό. Μπορεί να μας απαντήσει η Επιτροπή πώς θα υπολογίζεται οι άδειε για τα γονικά επιδόματα και τα γονικά επιδόματα για τις εργαζόμενες με συμβόλαια μηδενικών ορών. Ξέρω, θα πείτε πως αυτό έχει να κάνει με το εθνικό δικαίο και εθνικές πολιτικές. Ρωτάω όμως, δεν είναι αντιφατικό από τη μια να ισχυρίζεται η Επιτροπή πως με την πρόταση αυτή θέλει να βοηθήσει στην ρύθμιση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και από την άλλη να κλείνει τα μάτια μπροστά στην απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Γιατί όπως μπορεί να σερωπήσει κανείς την προσωπική του ζωή όταν έχει πλήρως απορριθμιστεί η επαγγελματική του ζωή. Επίσης, μπορείτε να μας πείτε γιατί η διάρκεια της άδεια πατρότητας δεν είναι ίδια με τη διάρκεια της άδεια μητρότητας τουλάχιστον. Και προσοχή, μην με την άδεια μητρότητας και την άδεια λοχίας, που είναι κάτι που αφορά μόνο την μητέρα, έχει να κάνει με την αποκατάστασή της. Και άλλο ένα θέμα στο οποίο δεν άκουσα να αναφέρεστε. Τι γίνεται με τις μονογονεϊκές οικογένειες. Δεν υπάρχει καν αφορά στο κείμενο της πρότασης σε αυτές. Δεν νομίζετε ότι η ευάλωτη αυτή κατηγορία του πληθυσμού πρέπει να χαίρει επιπλέον προστασίας. Το ανέφερε πριν και ήταν Γκονζάλες. Το ίδιο ισχύει και για τους γονείς με αναπηρίες. Έχει κάποια πρόταση η Κομισιόν σχετικά με αυτό. Τέλος, μπορεί να μας πει τι εννοεί η Επιτροπή ως επαρκές επίδομα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 της πρότασης. Επαρκές με κριτήρια μισθών Λουξεμβούργου ή μισθών Βουλγαρίας. Σταματάω εδώ και σε ευχαριστώ. Ε, ε, ευχαριστούμε. Ορτασούν. Δεν είναι εδώ. Ντανιέλα Γιούτο. Ούτε. Μιλένα Τροσίσκι, Ούτε. Ούτε. Αυτό σημαίνει ότι περάμε στο κατάλογο ομιλητών. Η κυρία Γιονγκέριους λοιπόν πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπα και πριν, τρία πράγματα θέλω να ρωτήσω για την πρόταση αυτή. Πρώτον, η πρόταση η ίδια μιλάει για αμοιβόμενη άδεια σε επίπεδα αναρωτικής. Ερώτηση εδώ, ερωτηματικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ποιος πληρώνει αυτή την αμοιβή. Γιατί στη χώρα μου, για παράδειγμα, η αναρωτική τα πρώτα δύο χρόνια της ασθένειας πέφτει στους ώμους των εργοδοτών, στην Ολλανδία τουλάχιστον έτσι είναι. Οπότε λένε γιατί να ξαναπληρώσουν. Οπότε, τι να υποθέσω, ότι από τη δικιά σας την πλευρά μιλάτε για το επίπεδο πληρωμής, αλλά όχι το ποιος θα πληρώσει. Μπορεί δηλαδή η συλλογική κοινωνική προστασία να πληρώνει, έτσι. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερον, μπορείτε να προβλέψετε πώς θα ανταποκριθεί το Συμβούλιο σε αυτή την πρόταση. Γιατί εμεί ακούμε διάφορα ανησυχητικά για χώρες μέλη που συνασπίζονται, δεν ξέρω εγώ πώς, Μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό. Και τρίτον, αν υπάρξει επιτυχία εδώ, θα κάνετε προτάσεις και για την άδεια μητρότητας. Πρόεδρος. Κύριε Μαρτάν, εσύ σκάνατε ήδη τις ερωτήσεις σωστά γιατί βλέπω εδώ το όνομά σας, αλλά υποθέτω δεν θέλετε να πάρετε πάλι το λόγο. Ωραία. Ωραία, τέλειωσε αυτός ο κατάλογος. Σόντροβα. Α, εδώ, ναι, ναι, σωστά, υπήρχε και η κυρία Σόντροβα. Συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο και θα είμαι σύντομη, γιατί θεωρώ ότι η πρόταση αυτή καθ' αυτή είναι πολύ θετική και πρέπει και φαντάζομαι ότι πραγματικά θα βοηθήσει να πετύχουμε αυτή την ισορροπία οικογενειακής και προσωπικής ζωής και επαγγελματικής ζωής, συγγνώμη. Το θέμα των 10 ημερών είναι πολύ φιλόδοξο για την πατρική άδεια. Εμείς έχουμε 5 μέρες στην Τσεχία με ένα σωρό προβλήματα. Οπότε η φιλοδοξία αυτή είναι πολύ απαιτητική κατά τη γνώμη μου. Είναι όμως μια καλή πρόθεση. Τέσσερις μήνες γονική άδεια που δεν μεταβιβιάζονται επίση, Πιστεύω ότι είναι μια σωστή κατεύθυνση για τα 12 πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού. Και η άδεια για όσους φροντίζουν οικείους επίσης. Τώρα για την ευελιξία ή μειωμένο ωράριο πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμο για τους γονείς μικρών παιδιών. Χαίρομαι επίσης και για την παράγραφο 8, την εγγύηση που αναφέρεται εκεί για μια κατάλληλη αμοιβή. Οι χώρες μέλη πρέπει να ξέρουν ότι δεν πρόκειται για μια συμβολική αμοιβή, αλλά για μια αμοιβή η οποία συνδέεται με τη συνεισφορά στο Ταμείο Ασφάλειας. πρέπει να δούμε ποιος τελικά ε, θα πληρώσει για αυτές τις αποφάσεις. Και για τους κοινωνικούς εταίρους και τα συνδικάτα έχω μια ερώτηση. Στην Τσεχία, όταν θέλαμε να εισάγουμε την ιδέα του home office, τα συνδικάτα δεν θέλανε να μπορεί ο εργαζόμενος να δουλεύει από το σπίτι του. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα πολύ καλό μέτρο και χαίρομαι που συμπεριλαμβάνεται εδώ. Ξέρω ότι με τους κοινωνικούς εταίρους, τα συνδικάτα θα υπάρξουν εντάσεις. Λυπάμαι όμως που τα συνδικάτα το αρνούνται αυτό, κυρίως τώρα που πρόκειται για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, και εγώ θέλω να πω δύο λόγια, επιτρέψτε μου. Είμαι από τη Σουηδία είμαστε γνωστοί για καλό σύστημα γονικής άδειας. Όταν συζητάμε στις Βρυξέλλες ή στη Σουηδία οπουδήποτε, μερικές φορές ακούω από τους εργοδότες ότι δεν συμφωνούν γιατί δεν υπάρχουν οικονομικά κέρδη από ένα τέτοιο σύστημα. Για μένα είναι πολύ κοντόφθαλμη αυτή η προσέγγιση. Γιατί η γονική άδεια μπορεί να μην έχει θετικές επιπτώσεις στα τρίμηνα των επιχειρήσεων, αλλά μακροπρόθεσμα για τις επιχειρήσεις είναι κάτι θετικό γιατί οι γυναίκες μένουν στην ε, αγορά, δεχάνουν χάνουν δεξιοτεχνίες κλπ. Και οι σύγχρονες επιχειρήσεις το γνωρίζουν αυτό. Και η Επίτροπος Γιούροβα το είπε όταν παρουσίασε την πρόταση αυτή. Επιχειρήσεις όπως η IKEA, για παράδειγμα, στηρίζουν τη γονική άδεια. Και να Μεγάλο μέρος της ε, ισχύω της ειδικής οικονομίας είναι ακριβώς αυτό, ότι φροντίζουμε για τις γυναίκες και για τους άντρες να μπορούν να συνδυάσουν την προσωπική με την επαγγελματική ζωή. Και όσο κερδίζουμε σε ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τόσο κερδίζουμε και σε ΑΕΠ, γιατί πρόκειται ουσιαστικά για επένδυση. Άρα είναι και οικονομικό το επιχείρημα και ελπίζω ότι δεν θα ακούσουμε και εδώ το αρνητικό επιχείρημα ότι δεν υπάρχει οικονομικό κέρδος. Και έπειτα ε, και οι πατεράδες ε, θέλουν να περνούν χρόνο με τα παιδιά τους όπως θέλουν και τα παιδιά τους ε, πατεράδες τους. Ήμουνα 44 όταν έκανα τη δεύτερη κόρη μου και ήμουνα υπουργό στη Σουδική κυβέρνηση. μια είναι μια χαρά και ο άντρας μου και τώρα δουλεύω πολύ σκληρά όπως δουλεύουμε όλοι. Οπότε ας περιοριστούμε στα στοιχεία, στα γεγονότα και όχι επειδή πρόκειται για άντρες, γυναίκες, οικογένειες, παραδόσεις. Να μιλάμε για την ισορροπία αυτή με έναν αξιοπρεπή και όριμο τρόπο. Έτσι πρέπει να κάνουμε πολιτική. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και τους άντρες και τις γυναίκες και τις οικογένειες. Καλώς. Τώρα, πολλές ήταν οι ερωτήσεις που ακούστηκαν. Οπότε έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Thank you very much. Um, Ευχαριστώ, προ... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ για τις τοποθετήσεις, τις ε, διάφορες ιδέες. Θα προσπαθήσω να κάνω και εγώ κάποια σχόλια. Και εφόσον θέλουν και οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση Just μπορούν να συμπληρώσουν. Είναι πολύ ενδιαφέρον ε, που ακούμε στις συζητήσεις σας ότι υπάρχει ευρεία συνένεση ότι υπάρχει δυσκολία. Υπάρχουν φραγμοί. Αυτό ακριβώ θέλει να αντιμετωπίσει η πρωτοβουλία, την εκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασία. Υπάρχει ανάγκη δράση. Κανεί δεν το αμφισβήτησε αυτό. Έχουμε μια σειρά από προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε από τη σκοπιά της απασχόλησης. Βλέπουμε κάποιες θετικέ τάσεις και βλέπουμε και οι άντρες να λαμβάνουν όλο ένα και περισσότερες ευθύνες προτιμώντα τι εργασιακέ διευθυντήσει που του επιτρέπουν να καλύψουν τι οικογενειακέ του υποχρεώσει. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αυτό το φιλόδοξο πακέτο για την εξισορρόπηση επαγγελματικού ιδιωτικού βίου, που ξεπερνά τα όρια απλώ τη άδεια μητρότητα και τη γονική άδεια. Γι' αυτό συμπεριλάβαμε και κάποια μη νομοθετικά εργαλεία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμιστεί. Ιδίω ό,τι αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας, είτε είναι φροντίδα παιδιού είτε άλλου μέλου τη οικογένεια, μέρο τη προσέγγιση που αναπτύσσει η ανακοίνωση για τη συμπλήρωση των κινήτρων από άλλους τομεί. Πάντως, πρόκειται για επένδυση. Επένδυση που μπορούμε να μεταφράσουμε σε ωφελήματα για τους γονείς, για τα παιδιά, για να υπάρχει καλύτερη κατανομή των υποχρεώσεων του επαγγελματικού και του ιδιωτικού βίου. Αυτά μπορούν να μεταφραστούν αυτομάτως σε υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης. Αυτό περιμένουμε από αυτά τα μέτρα. Αυτό από τις ε, εργασιακές συμβάσεις ή το όφελος που θα αποκομίσουν οι εταιρείε θα έχουν ίσως καλύτερα ποσοστά παραγωγικότητας καλύτερο συνδυασμό της ευελιξίας στην εργασία. Επίσης και θετικός αντίκτυπος στους ε, κρατικούς προπολογισμού. Όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα, το βραχυπρόθεσμο κόστος, το οποίο ε, βαθμία θα αυξάνεται οι χώρες που προέβλεψαν τα σχετικά μέτρα ε, σε ένα μεγαλύτερο φάσμα δεν τα αντιμετώπισαν όλα από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως ε, είναι αρμοδιότητα των 100 μελών να σχεδιάσουν ε, τη χρηματοδότηση των συστημάτων τους. Δεν είναι κάτι που θα το καθορίσουμε εμείς. Και δύο κουβέντες, γιατί αναφέρατε και κάποια άλλα ζητήματα, για το κατά πόσον θα μπορούν να μεταβιβαστούν τα δικαιώματα και για το κατά πόσον είναι εύστοχα. Αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της πρωτοβουλίας. Είναι πολύ σημαντικό και περιμένουμε να δούμε κάποιες θετικές προοπτικές απασχόλησης. Ιδίως ως προς τον απότερο αντίκτυπο. Για το κατά πόσον μπορούν να μεταφερθούν τα δικαιώματα ή όχι, μπορεί να το αποφασίσει η οικογένεια ποιο θα υποφεληθεί ή όχι. Τι είναι μεταβιβάσιμο και τι όχι. Εμεί θα σεβαστούμε την, το δικαίωμα επιλογή τη οικογένεια να αποφασίσει ή όχι. και μπορούν να την κάνουν την επιλογή τη στιγμή που θα περιμένουν το παιδί στην ε, αιστεία τους. Ε, για τους φροντιστές, όταν σε μια οικογένεια υπάρχει φροντιστής, Ιδίω όταν υπάρχει υποκατάσταση των επίσημων αναγκών ε, φροντίδας, της επίσημης υποχρέωσης φροντίδας, με μακροπρόθεσμη φροντίδα, είναι σημαντικό να το λάβουμε υπόψη. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους, Πιστεύω ότι η δέσμη αυτή μέτρων θα φέρει θετικέ αλλαγέ στα κράτη-μέλη προ καλύτερη εξισορρόπηση επαγγελματικού ιδιωτικού βίου και για να καλυφθούν τα χάσματα που υπάρχουν ή εναπομείνασε δυσκολίε. Ευχαριστώ. Απλώς να προσθέσω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με όσα υπόθηκαν σήμερα εδώ. Πρώτα απ' όλα, ένα σημείο που το θέξατε κι εσείς κύριε Σιγητά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς πρέπει να εξισορροπήσουμε όσα προτείνονται με τις υπηρεσίες και τι ευέλικτε διευθετήσει εργασία που μπορούν να προσφέρονται. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό στη συγκεκριμένη πρόταση και εδώ ε, βασιζόμαστε στο εξή ε, ιστορικό. Στι κοινωνίε μα ε, ο πληθυσμό γυράσκει. Έχουμε χαμηλά ποσοστά γεννησιμότητα γεννήσεων δηλαδή, και αυτό ε, ασκεί πιέσει στην αγορά εργασίας, είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό η συγκεκριμένη πρόταση δεν νομίζουμε ότι φύγει δυσανάλογα τις μικρομεσαίες. Ε, πρόσφατα στις εφημερίδες του Βελγίου διαβάσαμε ότι μεγάλες ε, εταιρείε όπως η Microsoft, η AXA, η ασφαλιστική έχουν διευθετήσεις πάνω από όσα προτείνει ο νόμος. Διότι ξέρουν τι κάνουν, θέλουν να διατηρήσουν τους εργαζόμενούς τους και γι' αυτό τους προσφέρουν κίνητρα. Και δεύτερον, αυτό ήταν το πρώτο. Εάν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στις προτάσεις αυτές, πρέπει να καλύψουμε και τις μικρομεσαίες. Σήμερα στην Ευρώπη είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας απασχολούν 80% του εργατικού πληθυσμού. Εάν τις αφήσουμε εκτός, χάνουμε τελείως το στόχο μας. Είναι λοιπόν προς το δικό μας το συμφέρον και των μικρομεσαίων υπό το φως της ε, μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας αυτοί οι κανόνες να ισχύουν και για εκείνες. Ιδάλλως τι θα κάναμε, πού θα παίρναμε την αγορά το εργατικό δυναμικό, Λόγω των δημογραφικών εξελίξεων έχουμε δύο επιλογές. τη μετανάστευση ή αξιοποιούμε όσο το δυνατόν περισσότερο το εργατικό δυναμικό που έχουμε. Έχουμε όμως πληθυσμό που στο ίμιση του έχει τεράστια προσόντα. Μπορεί να αξιοποιηθεί στον ύψιστο δυνατό βαθμό. Αλλά μακροπρόθεσμα οφείλουμε να σκεφτούμε τις μικρομεσαίες, διότι δεν απέχει και πολύ και αυτή η ανάγκη. Ποιος θα αντιμετωπίσει το κόστος που μπορεί να προκύψει. Εντάξει, όντω, και πρέπει να το διευκρινίσω και απαντώ έτσι και στην ερώτηση της κυρίας Γιονγκέριος. Η πρότασή μας δεν εξηγεί καθόλου αν το κόστος πρέπει να το αναλάβουν οι εταιρείε ή όχι οι ίδιες. Υπάρχουν ε, διαφορές μεταξύ των κρατών για το πώς το κόστος της κοινωνικής προστασίας ε, καλύπτεται ή όχι. Στην οδηγία λοιπόν τι κάνουμε, ορίζουμε ένα επίπεδο, ένα επίπεδο που ισχύει σε εθνική κλίμακα, ε, στο επίπεδο της ανερωτικής. Δεν διακδικάζουμε εμείς όμως ποιος θα πληρώνει. Υπάρχουν κάτι μέλη που οι άδειε είναι αμοιβόμενες. Εκεί πρέπει να βρεθεί σωστή ισορροπία μεταξύ του ότι καλύπτεται από τους εργοδότες και από την κοινωνική ασφάλεια. Πάντως, όταν οι άδειε αυτές είναι μεγαλύτερες διάρκειας όπως η γονική, δεν μιλάμε για τις πιο σύντομες, αυτές δεν πληρώνονται στο 100% από τι εταιρείε. Ίσως να υπάρχει λοιπόν προσδοκία ε, όταν ένα κράτο μέλο μεταφέρει την οδηγία αυτή σε εθνική νομοθεσία να εξισορροπήσει, να βρείτε λοιπόν το σωστό σημείο ισορροπία εθνική ε, κλίμακα για το τι πρέπει να πληρώνεται από τι εταιρείε και τι όχι. Από τον ε, κρατικό κορβανά. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό. Η οδηγία δεν λέει. Δεν λέει ποιο θα πληρώνει τι. Κατά δεύτερον, ποιο είναι αυτό το κόστος πέραν της κάλυψης του κόστους της άδεια ή διοργάνωση της υποκατάστασης λόγω χάρη. Πρέπει να αντικατασταθεί ένας εργαζόμενος που θα σε άδεια. Πρέπει να διοργανωθεί εν μέρη το φόρτος εργασίας στη, στη δουλειά. Εκεί κοιτάζουμε λοιπόν να υπάρχει όσο δυνατόν λιγότερος φόρτος. Ας πούμε με τη γονική άδεια. Δίνουμε τη δυνατότητα σε εταιρείε να πούν όταν ένας εργαζόμενος ζητά άδεια, μπορείτε να πείτε δεν είναι ακόμα κατάλληλη στιγμή, έχουμε κάποιες δυσκολίες στη λειτουργία της επιχείρησης, πάρτε μετά την άδεια. Οι εργοδότες μπορούν να αναβάλουν τη γονική άδεια. Υπάρχει δυνατότητα όταν ένας εργαζόμενος ζητά ελαστικές ε, διευθετήσεις να υπάρξει άρνηση και να του πει ο εργοδότης «Α, δεν γίνεται τώρα, δεν βολεύει, εάν κάθε πρωί πρέπει να υπάρχει κάποιο λόγου χάρη για να κάνει για να κάνει κάποια δουλειά σε ένα γκισέ, μπορεί ίσως να μην μπορεί μια μικροεπιχείρηση να πει φύγε με άδεια, όποτε θες. Ο εργοδότης μπορεί να αρνηθεί αν δεν βολεύει. Δεν ταιριάζει με το σύστημα ή το, τον τύπο διοργάνωσης της εταιρείας. Εάν υπάρξει πάντως τέτοια αρνητική απάντηση, δεν χρειάζεται να είναι γραπτή. Έχουμε πει πολλά που δείχνουμε ότι προσέχουμε και το σκέλος των εργοδοτών. Διαβάστε με προσοχή όλες τις διατάξεις και αν υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ελάφρυνσης και να το δούμε. Πάντως, κάναμε όσο πιο light γίνεται τις διατάξεις. Αυτό ήταν το πρώτο για τις μικρομεσαίες. Επίσης ακούστηκε, αλλά δεν είμαι βεβαία, νομίζω η κυρία Κοσλόφσκα το είπε, ότι σήμερα σε αρκετά κράτη-μέλη υπάρχει ένα συνολικό πακέτο αδειών για την οικογένεια και η οικογένεια επιλέγει πώς θα τις ε, ε, χρησιμοποιήσει. Πώς θα ασκήσει τα σχετικά δικαιώματα. Δεν θέλουμε να μειώσουμε αυτή την ευελιξία, να την περιορίσουμε. Όμως το να υπάρχει ε, μια περίοδος μη μεταβιβάσιμη για τον πατέρα έχει κάποια διαφορά. Διότι στα συστήματα όπου οι οικογένειες είναι ελεύθερες ε, να επιλέγουν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, η οικογένεια δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της, αυτός που βγάζει τα περισσότερα λεφτά στην οικογένεια, να πάρει άδεια, διότι χάνεται ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματο. Άρα συνήθως είναι ο ε, δεύτερος που σε ε, τιμές κερδίζει εισόδημα για την οικογένεια, η μητέρα δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι λίγο απογοητευτικό που με τη συζήτηση αναφερόμαστε στην ε, ευελιξία για τις οικογένειες, το ότι κάνουν ό,τι θέλουν και επιλέγουν ελεύθερα. Δεν είναι έτσι. Συνήθως οι μητέρε παίρνουν την άδεια. Γι' αυτό λοιπόν προβλέπουμε αυτή την περίοδο ειδικά για τους πατέρες, για να έχουν αυτό το εξατομικευμένο δικαίωμα που δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ε, για άδεια. Δεν μπορούν να το μεταφέρουν σε άλλον. Και τέλος, τέθηκε μια ερώτηση για το αν είμαστε εφόσον υπήρξαμε επιτυχεί ω τώρα, γιατί θέλουμε να θεωρήσει τι οδηγίε τη άδεια μητρότητα. Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί, εξηγήθηκε από την κυρία Αρένα, μετά το αδιέξοδο, το τέλμα στο οποίο περιλήφθαν οι συζητήσει για την άδεια μητρότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα σύνολο μέτρων για όλη την οικογένεια, αυτό συμβαίνει τώρα, και Προ δεν προβλέπουμε αναθεώρηση τη οδηγία για την άδεια μετρότητα, διότι θεωρούμε ότι οι συζητήσει ήδη εξέφρασαν την ε, πραγματικότητα οι περισσότερες εγγυήσει και διασφαλίσεις υπάρχουν. Τώρα μας ενδιαφέρει η υλοποίηση αυτών των εγγύησεων. Γι' αυτό στην ανακοίνωση για την εξισορρόπηση έχουμε μια συγκεκριμένη δράση. Σκοπό έχει να βελτιώσει την εφαρμογή και την άσκηση των υπαρχόντων δικαιωμάτων τη άδειας μητρότητας. Αυτό θα γίνει φέτος. Οργανώσαμε ενό είδου σεμινάριο εργαστήριο, όπω όπως θέλετε πείτε το, με ε, παρατηρητήρια των αγορών εργασία των διαφόρων κρατών για να δούμε πώ τα δικαιώματα αυτά θα ασκηθούν καλύτερα στο μέλλον. Ω προ το πώ θα τοποθετηθεί το Συμβούλιο και τι θα γίνει εκεί, ρωτήσατε από την Προεδρία. Γίνονται εκεί συζητήσεις ε, όπως και αυτές που γίνονται εδώ, μη μεταφορά, ε, αμοιβή, μηχανισμός για τους φροντιστές και σχετική άδεια, όλα αυτά συζητιόνται. Και υπάρχουν κάποιες χώρες με παρόμοιες απόψεις που συμπαρατάσσονται, ελπίζουμε να πετύχει να έχουν όλη την ίδια άποψη η Βουλγαρική Προεδρία. Είναι πολύ φιλόδοξη για το θέμα αυτό. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα οδηγήσει και σε κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ όλες και όλους, λέει η Πρόεδρος κυρία Ουλφσκόγκ. Εσείς κύριε Μαρτάν θέλετε κάτι να προσθέσετε. Ορίστε. Δεν ξέρω αν μπορεί να επανέλθει κανείς γιατί αυτά που μας είπατε είναι στην ουσία ο τετραγωνισμός του κύκλου ε, και ποιο ξέρω αν ποιος θα πληρώσει και αν δεν είναι η επιχείρηση τότε θα είναι τα δημόσια οικονομικά. Επανέρχεστε σε αυτό που ρώτησε η κυρία Γιονγκέριους. Τώρα καταλαβαίνω και λίγο καλύτερα γιατί υπάρχει αυτό το μπλοκάρισμα και βέβαια φαίνεται και από τη Γαλλία. Δεν εντυπωσιάζομαι διότι όλες οι χώρες μέλη έχουν κάνει νομικές ρυθμίσεις για να μειώσουν το κόστος της εργασίας η οδηγία για την συμφιλίωση του προσωπικού και επαγγελματικού βίου, ε, μα δεν θα δεχθούν να αυξήσει ξαφνικά πάλι το κόστος της εργασίας. Υπάρχουν ε, χώρες, ε, χώρες μέλη οι οποίες είναι όλες στο μείον. Κανείς δεν μπορεί να επενδύσει. Αν λοιπόν δεν είναι οι εργοδότες και αν δεν είναι ούτε τα δημόσια, τα δημόσια οικονομικά, ποιος θα, ποιος θα πληρώσει. Τελικώς ο κίνδυνος είναι θα πληρώσει ο ή η μισθωτή. Ο μισθωτός αυτός μπορεί να είναι ο κίνδυνος να πει «Α, ναι, λέτε, θα προτιμήσει να απαρατηθεί αν έχει τη δυνατότητα ή να κάνει κάτι άλλο». Πάτε λοιπόν επιτέλους, να, ξαναλέω, να τετραγωνίσει τον κύκλο με διαβήτη και κανόνα. Τι θα κάνετε, πρέπει να φανεί ε, θαραλέα και επιθετική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει όποιοι ε, όποιες χώρες χρηματοδοτήσουν από τον δημόσιο προϋπολογισμό να τους ε, υπολογιστεί διαφορετικά το δημόσιο έλλειμμα. Αλλά δεν το έχετε κάνει αυτό. Θέλετε να προσπαθήσετε να απαντήσετε στην ερώτηση του κ. Μαρτέν. Yes, thank you. Ναι, σας ευχαριστώ. Ε, ε, βεβαίως, τα χρήματα από κάπου θα πρέπει να προέλθουν και είναι σαφές αυτό βεβαίω θα ξεκαθαριστεί στο εθνικό επίπεδο εάν θα είναι ο δημόσιο προπολογισμό ή αν θα είναι ιδιωτικές επιχειρήσει. Συνήθω για μακροχρόνιε άδειε, συνήθω είναι ο προπολογισμό. είναι δηλαδή το δημόσιο το οποίο πληρώνει αυτό που θέλουμε εμεί να εξετάσουμε. όπω είπε και η πρόεδρο. το ζήτημα δεν είναι να το δούμε ω θέμα κόστου, αλλά ω επένδυση. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στην μελέτη αντικτύπου. Αποδείχνουμε ότι μακροπρόθεσμα θα έχει ευεργετική επίδραση στο ΑΕΠ και επομένως και στα δημόσια οικονομικά. Βέβαια, να μου επιτρέψετε να προσθέσω το εξή, λέει ο εκπρόσωπο τη άλλη Γενική Έχω κάποια εμπειρία σχετικά. Αυτά δεν γίνονται μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορείτε να πάτε από το 0 στο 30 στο 50%. Αυτή η ανάλυση κόστους κόστους-οφέλους πρέπει να μπει σε μια πιο δυναμική προοπτική. Υπάρχουν αλλαγές που καμιά φορά χρειάζονται χρόνο για να επέλθουν. Και η ρύθμιση που προβλέπουμε εμείς εδώ είναι σταδιακή. Ε. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Εδώ έληξε η συνεδρίαση. Βεβαίως παραμένουν πολλές ερωτήσεις. Ορισμένοι Κάποιοι θα απαντήσουν στην απάντησή σου, Μαρτέν, με φόροι. Οι φόροι θα πληρώσουν αυτά τα πράγματα. Όσοι έχουν υψηλούς μισθούς θα πληρώσουν υψηλότερου φόρους και αυτοί που έχουν χαμηλό εισόδημα δεν θα πληρώσουν τόσο πολλά. Αλλά αυτά σημαίνει δόμηση κοινωνίας, ε. πολιτικά τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ πάντως, λέει η πρόεδρος Ολφ Σκόγκ, όλες και όλους για την συμμετοχή σας. Χαίρομαι που τόσο ε, πολλοί άριθμοι ευρωβουλευτές παρέμειναν μέχρι τέλους, και έληξε η συνεδρίασή μας με αυτή την ε, πραγματικά ξεκάθαρη έτσι, ε, συζήτηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας εδώ. Είμαι βεβαία ότι η συζήτηση αυτή δεν θα είναι και η τελευταία για το ίδιο αυτό το θέμα. Ευχαριστώ.